Ε, Καλημέρα σε όλους. Ξεκινάμε την συνεδρίασή μας, την πρωινή. Πρώτο σημείο της ημερήσιας διάταξης αφορά την υλοποίηση και λειτουργία των προοπτικών συστημάτων ραδιοπλοείας μέσω δορυφόρου. Ραδιοναυσιπλοείας. Έχουμε περίπου 30 λεπτά για αυτό το θέμα της ημερήσιας διάταξης ε, νομίζω ότι η οργάνωση αυτών των συζητήσεων ξεκινά από την παρουσίαση της εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του κυρίου Φλαμόμαν. Ε, με συγχωρέστε μας, αλλά είναι τεράστια αίθουσα και έτσι δεν μπορούμε να σας δούμε καλά. Θα σας δώσω αμέσω εγώ λοιπόν στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μια παρουσίαση του προγράμματος μετά στον συγητή Μαρινέσκου και μετά θα μιλήσουν εκείνοι που ζήτησαν το λόγο. Λοιπόν, ο κ. Φλαμό ξεκινάει, έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καλημέρα κυρίες και κύριοι βουλευτές. Θα είμαι σχετικά σύντομο στην παρουσίασή μου, έτσι θα επιτραπεί μια συζήτηση επί του θέματος και έτσι έχετε δυνατότητα να θέσετε και ερωτήσει. Καταρχάς, θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι αντιπρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Σταγιάννη, ήδη έκανε μια παρουσίαση σχετικά σύντομη της προτάσεως κανονισμού σε αυτή την Επιτροπή μετά την έγκρισή του από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πέρσι τον Νοέμβριο. Έκανε την παρουσίασή σας εδώ σε εσά αρχές Δεκεμβρίου για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτές οι στιγμές της οικονομικής κρίσης θεωρούμε ότι το σύστημα δορυφορικής αδιοπλοείας Γαλιλαίο και Έγνο είναι σημαντική συνεισφορά εξ 2020 για την οικονομική ανάπτυξη, για την ανταγωνιστικότητα επίσης και εμπεριέχει ε, πολλές δυνατότητες, μεγάλες δυνατότητες για ανάπτυξη εφαρμογών και για την δημιουργία θέσεων απασχόλησης στην Ευρώπη να πω κάποια πράγματα όσον αφορά την παρούσα κατάσταση και μετά θα έρθω στην πρόταση κανονισμού σε ένα λεπτό Καταρχάς επιθυμίσω ότι η ραδιοναυσιπλοή αποτελείται από αυτή τα δύο προγράμματα. Το πρώτο είναι το EGNOS, το οποίο βελτιώνει το σύστημα GPS πάνω από την Ευρώπη. Αυτό το σύστημα είναι λειτουργικό εδώ και δύο χρόνια. Λειτουργεί πολύ καλά. Είμαστε πολύ υπερήφανοι. Για μας αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι οι χρήστες αρχίζουν στην πράξη να χρησιμοποιούν το σύστημα και κυρίως η πολιτική αεροπορία αρχίζει να το χρησιμοποιεί διότι περίπου καμία εκατοστή διαδικασίας προσγείωσης σε πολλά αεροδρόμια στην Ευρώπη ξεκινά να χρησιμοποιούν αυτή τη διαδικασία που έχει πάρει πιστοποίηση. Το δεύτερο κομμάτι της ε, ναυσιοπλοείας είναι το Γαλιλαίος. 21 Οκτωβρίου ξεκινήσαμε, ε, ε, μάλλον εκτοξέσαμε τους δύο πρώτους δορυφόρους που λειτουργούν. Αυτοί οι δορυφόροι λειτουργούν ιδιαίτερα καλά και οι συνάδελφοι μας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος μας ενημερώνουν εβδομαδιαία και μας δείχνουν ότι αυτοί οι δορυφόροι πετυχαίνουν τις επιδόσεις για τις οποίες ε, σχεδιάστηκαν. Ε, θα διαβάσατε στον τύπο ότι στις 2 Φεβρουαρίου αποφασίσαμε να προχωρήσουμε επιταχύνοντας ακόμα περισσότερο την ανάπτυξη των υποδομών διότι αποφασίσαμε να δώσουμε και άλλες συμβάσεις για 8 νέους δορυφόρους ε, καθώς και συμβάσεις ε, που θα εξασφαλίσουν ότι εκτοξευτές, ο εκτοξευτής Αριάν 5 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εκτόξευση των δορυφόρων και τη θέση του τροχιά και αυτό θα γίνει συμπληρωματικά πέραν από τις πυράβλους ογιούς που εκτοξεύονται από την Ευρωπαϊκή ε, Βάση Κουρού στην Γαλλική Γουιάννα. Θα έχουμε τελικά 26 δορυφόρους τροχιά το 2015 και ήδη μπορούμε να έχουμε αρχικές υπηρεσίες που παρέχονται ε, αρχές του 2014. Όσον αφορά την πρόταση κανονισμού που τελεί αντικείμενο της σημερινής συζήτησης, αυτή η πρόταση κανονισμού καλύπτει όχι μόνο την ολοκλήρωση των υποδομών, αλλά εξίσου και την εκμετάλλευση από το 2014 με το 2020 των δύο υποδομών Έγνος και Γαλιλαίος. Η πρόταση κανονισμού εδράζεται επί πολλών εγγράφων και πολλών δραστηριοτήτων, ε, ε, μεταξύ των οποίων και η περσινή έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Υπεύθυνο ήταν και ο Γόμεκ. Ε, βασιζόμαστε και επί των συμπερασμάτων του Συμβουλίου Μεταφορών του περσινού έτους. Κάναμε ανάλυση συνεπειών και εξυπακούεται ότι βασιζόμαστε επί της εμπειρίας μιας δεκαετίας όσον αφορά τη σύναψη συμβάσεων και το πώς χειρίζεται η ΕΣΑ, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος, αυτές τις συμβάσεις. Η βασική αρχή που ακολουθούμε στον κανονισμό είναι απλώς ο καθορισμός των ευθυνών, σαφής καθορισμός και η εκ νέου χρήση εμφισμένων φορέων ή υποδομών. Δηλαδή η διαχείριση του προγράμματος θα ανατεθεί στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Genesis, η ΖΕΣΑ, που εδρεύει στην Πράγα, δημιουργείται στην Πράγα τώρα. Θα ξεκινήσει η υπηρεσία τη διαχείριση των υποδομών έγνος από 1η Πρώτου 2014 και ε, εξάλλου σταδιακά θα αναλάβει τις δραστηριότητες ε, διαχείρισης ε, του συστήματος Γαλιλαίος. Παράλληλα θα συνεχίσει την προετοιμασία της αγοράς για την ανάπτυξη εφαρμογών και την εμπορική διάθεση των εφαρμογών. Διότι εξυπακούεται ότι δεν είναι η δημιουργία των υποδομών που είναι αυτός σκοπός, αλλά πιο πολύ η χρήση και η διάθεση στους Ευρωπαίους πολίτες των συστημάτων ραδιοναυσιπλοείας για να μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυτές οι υπηρεσίες σε πολλές εφαρμογές. Όπως έλεγα βέβαια δεν θέλουμε να επαναλάβουμε τα εφιστάμενα μέσα, να τα επικαλύψουμε και γι' αυτό θα συνεχίσουμε τη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματο που έχει αποκτήσει τεχνογνωσία ούτω ώστε να μπορεί να κάνει τι αναγκαίε βιομηχανικέ εργασίε τι οποίε έχει αναλάβει. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή η ίδια θα παραμείνει υπεύθυνη για τα προγράμματα στο σύνολό του. Θα έχει και την εποπτεία, θα εγγυηθούμε επίση την ασφάλεια των συστημάτων και θα ενημερώνουμε τακτικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Αυτά όσον αφορά τη διακυβέρνηση, τη διαχείριση των προγραμμάτων, όσον αφορά τα οικονομικά των προγραμμάτων, όπως σας είπα βασίσαμε τα στοιχεία μας και του υπολογισμού μας επί των αναλύσεων των λεπτομερεστάτων που απορρέουν από συμβάσεις που ήδη υπάρχουν, από την εμπειρία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος και τα κράτη-μέλη έχουν συμμετάσχει στον όλο υπολογισμό, διότι κάποια κράτη-μέλη έχουν μεγάλη εμπειρία όσον αφορά τα διαστημικά συστήματα και συμπεράναμε ότι ο αναγκαίος προϋπολογισμός για να μπορούμε να ολοκληρώσουμε τις υποδομές και να τις χρησιμοποιήσουμε θα είναι ένα δισεκατομμύριο ευρώ το χρόνο κατά τα έτη 2014-2020. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να επισέθω σε περισσότερες λεπτομέρειες όσον αφορά την πρόταση του κανονισμού. Είμαστε βεβαίως στη διάθεσή σας για να απαντήσουμε σε όλες τις ερωτήσεις που ενδεχομένω ε, έχετε. Ευχαριστώ. Συνάθος Μαρινέσκου έχει το λόγο. <coughs> Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον εκπρόσωπό τη για την παρουσίαση που μα έκανε. Εκτιμώ τη συνεργασία ε, που είχαμε ως τώρα. Έχω δύο ερωτήσεις να θέσω, είπατε. Ότι το GSA πρόκειται να αναλάβει την ευθύνη για την διαχείριση του προγράμματος, για τη λειτουργία του προγράμματος και το, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος είναι επίσης εν μέρη αρμόδια. Θα ήθελα να διευκρινίσουμε πού βρίσκεται ακριβώς το όριο Ποιε είναι ακριβώς οι αρμοδιότητε του GSA και ποιε είναι ακριβώς οι αρμοδιότητε του ESA, της Ευρωπαϊκής ε, Υπηρεσία για το Διάστημα και πώς μπορούμε να εξαλείψουμε την πιθανότητα σύγχυση. Επίσης, να ζητήσω από τον εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θεωρεί ότι υπάρχει σύνδεση μεταξύ του έργου αυτού και της χρήσης του για μελλοντικές εφαρμογές. Ευχαριστώ. Ε, Σας ευχαριστώ. Νομίζω ότι πρώτα θα ακούσουμε και άλλες ερωτήσεις και μετά θα δώσουμε το λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σίλβια Τσικάου, όλ, και μετά ακολουθούν οι επόμενοι. Thank you, Madam Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι θα πρέπει να καλωσορίσουμε τον κανονισμό που έχουμε μπροστά μας σήμερα και γι' αυτό για μια σειρά λόγων. Καταρχάς είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρξει μια μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση και διαχείριση αν θέλουμε να επιτύχουν τα προγράμματα Γαλιλαίο και Έγνος. Κατά δεύτερον, νομίζω ότι μπορούμε να καλωσορίσουμε τον κανονισμό αυτό γιατί είναι κρίσιμο τα προγράμματα αυτά να παραμείνουν πραγματικά ανεξάρτητα και να διασφαλιστεί ότι όλα τα κρατή-μέλη έχουν ίση πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές. Είναι σημαντικό λοιπόν το ότι ο κανονισμός διευκρινίζει ότι η Ένωση είναι ο ιδιοκτήτης των συστημάτων έγνωσης και γαλιλαίων και κατά τρίτον, Νομίζω ότι είναι σημαντικό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να έχει σημαντικό ρόλο επισκόπησης για να διασφαλίσει την καλύτερη λογοδοσία και διαφάνεια. Ελπίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει διδαχτεί από τις παρόμοιες δυσκολίες που έχουμε αντιμετωπίσει στο παρελθόν σε ό,τι αφορά παρόμοια προγράμματα. Νομίζω ότι υπάρχουν ε, το δίχως άλλος κάποια ζητήματα τα οποία πρέπει να διευκρινιστούν περαιτέρω. Για παράδειγμα, στην περίοδο 2014 και 2020 σε ό,τι αφορά ε, το Γαλιλαίο. Αυτό δεν περιλαμβάνεται απαραίτητα στις διαπραγματεύσεις, αλλά στις διαπραγματεύσεις για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Αλλά το θέμα ε, του πλεονάσματος των υπερβολικών εξόδων επίσης ε, θα πρέπει να το κοιτάξω. Έχουμε 7,9 δισεκατομμύρια ευρώ, προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι διπλασιασμός και πλέον της, του τρέχοντος ποσού, αλλά δεν προκύπτει από κάπου το πώς υπολογίστηκε το ποσό αυτό. Άρα θα μπορούσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας πει πώς κατέληξε στο ποσό αυτό. Είναι σαφές ότι θα πρέπει να διασφαλίσουμε στο μέλλον να μην υπάρχει ε, υπέρβαση του κόστους, γιατί στην περίπτωση αυτή υπάρχει κίνδυνος σε άλλα προγράμματα του ε, του κεφαλαίου 1α, όπως ο Horizon 2020, να διακυβευθούν αν ξεκινήσει τέτοιος ανταγωνισμός ε, για τους πόρους. Νομίζω ότι σημειώνεται πρόοδος για θέματα διαχείρισης και θα πρέπει πραγματικά να ασκήσουμε πίεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνεχίσει με πιο στεναρές δομές διαχείρισης και χαίρομαι που ελήφθη η απόφαση να διαγραφεί η πρόταση για τον κύκλο ζωής. Και τέλος, υπάρχει μία διάταξη για να ωφεληθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις από τα προγράμματα. Στην Επιτροπή μας ε, μας απασχολεί ιδιαίτερα το θέμα αυτό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, προκειμένου να λάβουν όσο πιο μεγάλη ενίσχυση γίνεται, γιατί ασφαλώς και αποτελούν βασική πηγή θέσεων εργασίας. Γι' αυτό λοιπόν είναι και τόσο σημαντικό το άρθρο 20. Ευχαριστώ. Και τώρα η Σιλβετικάο. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις πληροφορίες που μας έδωσε σήμερα το πρωί. Και έχω μία σειρά ερωτηματών, της απευθύνω. Σε ό,τι αφορά το άρθρο 14 14.1. Σύμφωνα με τον κανονισμό, τα συστήματα και η λειτουργία τους είναι ασφαλή. Αυτός ασφαλώς είναι ένας θεμητός στόχος, αλλά μία απλή δήλωση του γεγονότος αυτού δεν επαρκεί. Ιδιαίτερα κοιτώντα την παράγραφο 2 όπου αναφέρεται επιπροσθέτως ότι μέσω πράξεων κατά εξουσιοδότηση βάσει του άρθρου 34 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να υιοθετήσει προδιαγραφές για να εξασφαλίσει την ασφάλεια των ε, εγχειρημάτων που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Νομίζω ότι μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει κάπως να ε, βελτιώσουμε το κείμενο αυτό και το ίδιο ισχύει και για το άρθρο 13 οι διάφορες υπηρεσίες ε, λαμβάνουν διάφορες αρμοδιότητες σε ό,τι αφορά την ασφάλεια των προγραμμάτων. Το άρθρο 13.2d δέλτα αναφέρει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούσε να δώσει πιο πολλές ε, λεπτομέρειες σε ό,τι αφορά την ασφάλεια των προγραμμάτων. παρακολούθησα τα διάφορα στάδια ανάπτυξης των δύο προγραμμάτων Γαλιλαίου και Εγνός. Και στο πλαίσιο του προγράμματος Εγνός θα ήθελα να ρωτήσω πότε θα καλυφθεί το σύνολο της επικράτειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το πρόγραμμα. Από την παρουσίαση των προγραμμάτων ε, συναγάγω ότι το Γαλιλαίο θα καταστεί λειτουργικό σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση μόλις το 2020. Για τους ψηφιακούς ταχογράφους, για παράδειγμα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε μια διαφορετική πρόταση. Το πρόγραμμα GNSS ε, θα χρησιμοποιηθεί για τους ψηφιακούς ταχογράφους. Αυτή ήταν η πρόθεση, ωστόσο, αυτή η ψηφιακή ταχογράφη που θα χρησιμοποιούν τα σήματα GNSS θα πρέπει να καταστούν λειτουργικοί μέχρι το 2018. Διακρίνω λοιπόν μία αντίφαση στο σημείο αυτό σε ό,τι αφορά την χρονική συγκυρία. Αν το σύστημα θα καλύψει το σύνολο της επικράτησης Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2020, πώς θα καταστεί δυνατόν να προαπαιτηθεί το 2018 να χρησιμοποιούνται σε όλη την επικράτεια η ψηφιακή ταχογράφη. Θα μπορούσε να μας απαντήσει λεπτομερώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα ήθελα να συνεργαστούμε εντελεχώς σε ό,τι αφορά το θέμα της ε, κάλυψης της πανευρωπαϊκής. Γιατί δεν με ενδιαφέρει μόνο ε, ο δορυφόρος σε τροχιά και η βάση του θέλω να ισχύσει και για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και σε ό,τι αφορά κατά τι εφαρμογέ των συστημάτων, θεωρώ ότι είναι σημαντικό να μα διασφαλίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι το πρόγραμμα Horizon 2020 θα συμπεριλάβει την απαραίτητη χρηματοδότηση έρευνας για την ανάπτυξη εφαρμογών και υπηρεσιών που χρησιμοποιούνται από τα συστήματα Έγνος και Γαλιλαίου. Σύντομα θα υπάρχουν υποδομές ε, δορυφορικές ε, και οι ανάλογες, οι σταθμοί βάσης. Όλα αυτά καλά και ωραία, αλλά αν δεν υπάρχουν οι ανάλογες υπηρεσίες και εφαρμογές, το σύστημα πολύ απλά δεν θα χρησιμοποιηθεί για τον σκοπό για τον οποίο ε, συλλήφθη και δεν θα αξιοποιηθεί το δυναμικό του τελευταία ερώτηση σε ό,τι αφορά τη μελλοντική διαχείριση. Μέχρι το 2020 υπάρχει σαφές σχέδιο σε ό,τι αφορά την πρόταση του κανονισμού. Ερώτημα όμως προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ποιος θα είναι υπεύθυνο για το λειτουργικό τμήμα μετά το 2020. Ποιος θα είναι υπεύθυνο για τη χρηματοδότηση και ποιος θα είναι υπεύθυνο για τους ανθρώπινους πόρους. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Έχουμε αρκετούς εγγεγραμμένους για να πάρουν το λόγο. Έχουμε εξαντλήσει και το χρόνο για αυτό το θέμα. Και παρακαλώ, ξέρω ότι είναι σημαντικό το θέμα, αλλά παρακαλώ να είσαστε λίγο σύντομοι, αν έχετε την καλοσύνη. Ε, Κύριο Λαμπέρ, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Έχω δύο ερωτήσει και οι δύο ερωτήσει σχετίζονται με τον υπολογισμό. Είναι κάτι που δεν καταλαβαίνω πολύ καλά στο πρόγραμμα σχέδιο κανονισμού. Μιλάμε για 7 εκατομμύρια 7,8 δισεκατομμύρια. Είπατε ένα εκατομμύριο το χρόνο επί 7 κάνει 7 δις και λέτε 7,8. Μιλάμε για πλήρη εφαρμογή και ασφάλεια ή χωρίς safety of life με ή χωρίς safety of life safety of life. Αυτό είναι το πρώτο ερώτημα. Μιλάτε για περιθώριο σφάλματος. Γιατί στον προπολογισμό. Δεύτερο στοιχείο. Τι διαδρομές φτύλης μπορούμε να ακολουθήσουμε αν θέλουμε να επιτρέψουμε η στετιωτική χρήση του Γαλιλαίου να πληρώνεται από τα κράτη-μέλη. Σκεφτήκατε ποιες δυνατότητες είναι κομμάτι του προπολογισμού Γαλιλαίος να καλύπτεται από άμεση εισφορέ των κρατών μελών στο βαθμό της χρήση για τι υπηρεσίε ασφάλειας. Κάτι που δεν αφισβητούμε, όμως ο καθένας θα πρέπει να καταβάλει τα δικαίως οφειλόμενα. Ευχαριστώ. Το Τζενόσκι. Ο κύριος Τζενόσκι. Ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε. και εγώ να ευχαριστήσω την Επιτροπή για την φρέσκια αυτήν ενημέρωση. Να μην επαναλάβω αυτά τα οποία είπαν οι συνάδελφοι, ήταν πολύ χρήσιμο όσα είπαν και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ θετικό το ότι τώρα γνωρίζουμε πώς στην πράξη θα αξιοποιηθεί αυτή η υποδομή. Τώρα είναι ξεκάθαρο τι χρονοδιάγραμμα έχουμε όσον αφορά αυτούς τους δορυφόρους. Αυτό που εγώ θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό και συμφωνώ με αυτούς που το σχολίασαν είναι ότι τώρα έχουμε μια πιο ξεκαθαρή άποψη για το τι ισχύει και για τη χρηματοδότηση. Πρόκειται να εμφανιστούν εφαρμογές από διάφορους ευρωπαϊκούς φορείς όμως θα έχουμε και Παραμογές θα έχουμε και από πανεπιστήμια. Να δούμε επομένω πώς θα έχουμε κάποια ιδέα που είναι χρήσιμο. Να μας πει δηλαδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το τι είδους εφαρμογές ε, αναμένονται να εμφανιστούν στο μέλλον. Δεν θα τον περιμένει κανείς ούτε μέχρι το 2020 ούτε καν το 2014. Και πρέπει να δούμε επομένως τι γίνεται, πώ θα εξελίξουν ε, τα πανεπιστήμια αυτές τι εφαρμογέ που χρειάζονται κάποιο χρονικό περιθώριο για να μπορέσουν να τις εξελίξουν. Σας ευχαριστώ. Τελευταίος από του Σκιώδης, Ρέμεκ. Κύριος Ρέμεκ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε κυρία Πρόεδρε, και εγώ αισθάνομαι πάρα πολύ ικανοποιημένος μια που καταφέραμε να φτάσουμε σε αυτή την προχωρημένη φάση ε, της διαδικασίας για να αποκτήσουμε σχέδιο κανονισμού το κοινοβούλιο τώρα αποδεικνύει ότι επιτυχώς χειρίζεται τα σχετικά θέματα και στο μέλλον θα ισχύσει το ίδιο. Νομίζω ότι θα πρέπει να ε, φτιάξουμε έναν κανονισμό ο οποίος να υλοποιήσει όλα αυτά τα οποία οραματίζονται οι προηγούμενοι συνάδελφοι, όσοι μίλησα προηγουμένω. και επομένω θα πρέπει να αξιοποιηθούν κατά αυτόν τον τρόπο οι υπάρχοντες πόροι. Σε αυτόν τον ε, οργανισμό επίσης θα πρέπει να δούμε πώς θα εξασφαλίσουμε ανεξαρτησία και ευελιξία όσον αφορά για τους φορείς που θα χειριστούν αυτό το project. Η αλήθεια είναι ότι μα έχει ξαναπασχολήσει το θέμα αυτό, αλλά δεν έχουμε ακόμα ιδέα για το τι μορφή θα πάρουν αυτέ οι εφαρμογέ στο μέλλον. Αυτά και με μεγάλη μου χαρά θα συνεργαστώ με του υπόλοιπου συναδέλφου στο μέλλον. Νομίζω ότι θα πάνε τα πράγματα πάρα πολύ καλά. Σα ευχαριστώ. Δύο συνάδελφοι ζήτησαν να μιλήσουν, Βαν Ιστελρόι και Πρόντι. Κύριο κ. Βαν Ιστελρόι έχει το λόγο πρώτο. Ευχαριστώ πολύ. Έχω δύο σύντομε παρατηρήσει. Πρώτα πρώτα είναι πάρα πολύ θετικό το ότι προχωρούμε με γρήγορο ρυθμό συνεχώς και σοβαρά μας ενδιαφέρει επομένω το πώς θα διεκπαιρεώσουμε το θέμα για τον κανονισμό αυτό. Αυτή είναι η θέση του Κοινοβουλίου γιατί δεν έχουν πιστεί όλοι όσον αφορά τη χρηματοδότηση το τι θα γίνει. Επομένω, το ότι συνεχίζουμε την προσταθειά μα ε, αποτελεί ένα ξεκάθαρο μήνυμα το οποίο στέλνουμε. Κάτι άλλο τώρα ε, για βιομηχανία και για τη συμμετοχή. Θα πρέπει να θυμηθούμε το ότι τα πράγματα δεν πήγαν καθόλου καλά στην πρώτη φάση με τον Γαλιλαίο. Τι εγγύσει υπάρχουν ε, για την επόμενη φάση. Πολύ σημαντικό. Κάτι άλλο τώρα. Τι θα κάνουμε με τις τρίτες χώρες που θέλουν να χρησιμοποιήσουν τις εφαρμογές μας, τον εξοπλισμό μας, τις επενδύσεις μας, να δούμε τι συμβόλαια θα έχουν. Να δούμε. Έχουν τεθεί πολλές ε, ερωτήσεις και περιμένω και εγώ τις απαντήσεις. Ευχαριστώ Βιτόριο Πρόντι, ευχαριστώ Πρόεδρε. Συμφωνώ όσον αφορά τα υποθέτα. Όμως πρέπει να επιταχύνουμε τις επενδύσεις. Αν και για το Γαλιλαίος υπήρχαν και καθυστερήσεις και αυξήσεις των δαπανών. Αλλά αυτός δεν είναι σωστός λόγος για να αφήσουμε να χαθεί αυτό το πρόγραμμα, αλλά θα πρέπει να επιταχύνουμε, αντιθέτως. Και, και η οικονομική κρίση θα μπορούσε να είναι λόγος για να επενδύσουμε γρήγορα επ' αυτών των ευρωπαϊκών υποδομών. Μεταξύ άλλων θα πληρώσουν από μόνε τους αυτές οι υποδομές το κόστος τους. Θα ήθελα να πω ότι πρέπει να επιταχύνουμε όσο γίνεται διότι κάθε χρόνος κάθε, ο χρόνος που εξοικονομείται είναι χρόνος καύσιμο που εξοικονομείται κυρίως για τις ε, αερομεταφορές υπογραμμίζω ότι για όλους αυτούς τους δορυφόρους τους σχηματισμούς των δορυφόρων θα πρέπει να βρούμε τη σωστή θέση το ταχύτερο δυνατό πρέπει να εξοξευθούν και να τοποθετηθούν οι δορυφόροι. Και το GMS είναι σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό σύστημα και θα πληρώσει το κόστος του. Όλα αυτά θα έπρεπε να επαναξεταστούν. Και οι ευρωπαϊκές υποδομές θα πρέπει να είναι έτοιμες να δώσουν πλήρως τις υπηρεσίες τους ε, το ταχύτερο δυνατόν. Ευχαριστώ. Σιλβάνα Τσεκάου ζήτησε το λόγο. Το ζήτησε το λόγο Σιλβία, αλλά πάρα πολύ σύντομα, σε παρακαλώ. Σε ευχαριστώ, Πατρίτσια. Δοθέντος ότι τα δύο πρόγραμματα είναι προγράμματα πρώτης γραμμής για την Ευρωπαϊκή Ένωση και πολλοί τομείς της στην Ευρώπη εξαρτώνται από αυτά τα δύο προγράμματα. Θα συνέστηνα, κυρία Πρόεδρε και συνάδελφοι, να διοργανώσουμε μία συζήτηση, μία μίνι ακρόαση ενδεχομένω όσον αφορά τα προγράμματα Γαλιλαίος και Έγκνος και ίσως και το GMES και έτσι όλοι οι συνάδελφοι, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούσαν να σχηματίσουν σαφή εικόνα περί των ε, επιτευχθέντων και επί των μελουμένων και των δυνατοτήτων που θα, θα ε, παρουσιάσουν τα προγράμματα τα τρία στο μέλλον. Θα δούμε, οι συνάδελφοι του συζητάνε με του συντονιστέ και θα δούμε κατά πόσο αυτό είναι εφικτό, απαντάει η Πρόεδρο. Ο κ. Φλαμό έχει το λόγο, ε, γνωρίζοντα βέβαια ότι δέχτηκε πάρα πολλέ ερωτήσει. Λοιπόν, παρακαλώ στο βαθμό του δυνατού να είστε εξαντλητικό απαντήσει. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να απαντήσω στι ερωτήσει άνευ ε, χρόνου μετά ο επιμερισμό των ευθυνών μεταξύ Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματο και τη ε, Ευρωπαϊκή Αρχή του ZNSS, τη ZSA. Παίρνω το παράδειγμα του συστήματο EGNOS που είναι σχετικά απλό. Επί μία δεκαετία περίπου η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματο παρακολούθησε τεχνικέ εργασίε για τη σύλληψη και ανάπτυξη των υποδομών. Αυτοί, αυτές οι υποδομές λειτουργούν και σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χειρίζεται τις, τις διάφορες με τους διάφορους φορείς και χρήστες των δορυφορικών συστημάτων για την τοποθέτηση επίσης αντικειμένων που ήταν δορυφόρων και έχουμε και την προσωπή στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματο στο μέλλον. Αυτό ο ρόλο που κληρώνει σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εφαρμοστεί από την ΖΕΣΑ. Η διαφορά μεταξύ ΖΕΣΑ και τη Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματο. Ποια είναι, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματο για το σύστημα ΕΓΝΟΣ. θα ασχολείται με τι μελλοντικέ εξελίξει του συστήματο. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματο θα μα πει πώς να αλλάξουμε τα σήματα σε 5-10 χρόνια, πώς να βελτιώσουμε το σύστημα για να γίνει αποτελεσματικότερο, πώς να επικαιροποιηθεί, διότι όπως σας είπα το έγνος είναι ένα σύστημα που εδράζεται επί το GPS. Το GPS εξελισσόμενο σημαίνει ότι χρειάζεται και το έγνος να εξελιχθεί. Ε, εν συνέχεια, όσον αφορά τα 7 δις ευρώ και τη δυνατότητα να μην ξεπεράσουμε αυτό το κονδύλι, Κατά το παρελθόν πράγματι το σύστημα είχε κάποιες οικονομικές παρεκκλήσεις και θέλουμε να το αποφύγουμε αυτό. Στο μέλλον, όπως σας προανέφερα, τα στοιχεία τα οποία παρουσιάζεται σήμερα βασίζονται ε, επιφυσταμένων συμβάσεων, πραγματικών συμβάσεων. Ξέρουμε ακριβώς πόσο κοστίζει ένας δορυφόρο, πόσο ε, λειτουργεί ο φορέας που ελέγχει τον ε, δορυφόρο. Με βάση αυτόν αυτά τα στοιχεία επεξεργαστήκαμε τον προπολογισμό και στον προπολογισμό έχουμε βάλει και κάποιε προβλέψει για τον κίνδυνο διότι μεγάλα τεχνολογικά προγράμματα όπως αυτά δεν είναι προστατευμένα από προβλήματα τεχνικής φύσεω επίσης για να αποφύγουμε να πρέπει να επιστρέψουμε προς δημοσιονομικέ αρχές με αιτήματα για κονδύλια προβλέψαμε όπως γίνεται σε κάθε πρόγραμμα τεχνολογικό προθυμέ τεχνολογίας προβλέπουμε λέγω ένα απόθεμα σε περίπτωση προβλημάτων. Ε, συνεχεία όσον αφορά την ασφάλεια των συστημάτων. Ναι, στον κανονισμό εξηγούμε ότι τα συστήματα είναι ασφαλή. Για να μπορέσουμε να το πούμε αυτό, βασιζόμαστε επί κάποιων προδιαγραφών που περιλαμβάνουν απαιτήσει για την ασφάλεια. Αυτέ οι απαιτήσει για την ασφάλεια, οι προδιαγραφέ δεν εφευρίσκονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τι επεξεργάζονται τα κράτη-μέλη ε, που έχουν μεγάλη εμπειρία στον αφορά τη διαχείριση συστημάτων που χρειάζονται υψηλό επίπεδο ασφαλείας και τα κράτη-μέλη τα ίδια εκ των υστέρων ε, πιστοποιούν αυτά τα συστήματα για να είναι σίγουρα ότι τα συστήματα πληρούν τις προδιαγραφές τους. Το ότι περνούμε από κατεξισοδότηση πράξης, ε, αυτό το κάνουμε για λόγους νομικούς. Σε μία μήνυα ακρόαση ενδεχομένως θα μπορούσαμε να πούμε σε περισσότερες λεπτομέρειες. Όσον αφορά την κάλυψη του έγνος, ε, την κάλυψη της ευρωπαϊκής επικράτησης από το έγνος, ήδη καλύπτει μεγάλο κομμάτι της Ευρώπης το έγνος, αλλά κάποιες περιφερειακές ζώνες, όπως η Ανατολική Πολωνία ή οι Αζόρες, καλύπτονται λιγότερο καλά. Βεβαίως, βεβαίως προσπαθούμε να επεκτείνουμε την κάλυψη του έγνος σε όλη την Ευρωπαϊκή Επικράτεια και πέραν αυτής, διότι θέλουμε να καλύψουμε και την ΕΚΑΚ για την ε, πολιτική αεροπορία που συμπεριλαμβάνει περισσότερες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και θέλουμε ένα σχέδιο ανάπτυξης των διαφόρων σταθμών επί Ευρωπαϊκής Επικρατείας ούτω ώστε μακροπρόθεσμα να μπορέσουμε να καλύψουμε ακόμα και τις ε, περιφερειακές ζώνες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Όσον αφορά τους ψηφιακούς ταχογράφους, και, και πότε θα λειτουργεί 100% το Γαλιλαίος, αν θα λειτουργεί μέχρι το 2020. Το σύστημα ταχογράφων δεν θα βασίζεται μόνο αποκλειστικά επί των επιδόσεων του Γαλιλαίος και του Έγνος, αλλά εξίσου επί του Αμερικανικού συστήματος. Και οι συνάδελφοί μου, συνεπώς, που κάνουν τις προτάσεις για τους ταχογράφους, γνωρίζουν πολύ καλά ότι δεν θα βασιστούμε αποκλειστικά επί του Γαλιλαίου για να παράσχουμε αυτές τις υπηρεσίες. Όσον αφορά το σχεδιασμό μας. Μέχρι 2020 σχεδιάζουμε σήμερα. Βέβαια, επεξεργαζόμαστε και προβολές μελλοντικέ. Όσον αφορά τις ευθύνες των επιχειρήσεων και σηματοδοτήσεων, τη στιγμή που η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει αναπτύξει τις υποδομές και θέλει να λειτουργήσουν, οι δημόσιοι πόροι θα εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση της λειτουργίας του συστήματος και των συστημάτων όσον αφορά τη διαχείριση τις επιχειρήσεις, τη λειτουργία. Όπως είπαμε, η ΖΕΣΑ είναι η αρμόδια αρχή, η οποία μετά το 2020 θα διαχειρίζεται όλες τις ε, υποδομές. Για να απαντήσω στο ερώτημα για τα 7 δις ή 7,8 δις, τα 7 δις ευρώ αφορούν οικονομική κατάσταση του 2011, ενώ το 7,8 δις ή 7,9 δις είναι ένα στοιχείο που αντιστοιχεί στο σχέδιο ετησίων αναλήψεων υποχρεώσεων και λαμβάνει υπόψη και 2% πληθωρισμό το χρόνο. Όσον αφορά τη χρηματοδότηση από το στρατό τις στρατιωτικές αρχές, όταν θα χρησιμοποιήσουν οι στρατιωτικοί το σύστημα, το συζητούμε αυτό με τα κράτη-μέλη, όσον αφορά την χρήση PRS, και θέλουμε να δούμε κατά πόσο τα κράτη-μέλη που θέλουν να χρησιμοποιήσουν το PRS ε, θέλουν να πληρώσουν και δικαιώματα για τη χρήση του PRS ή όχι, αλλά δεν έχουν ολοκληρωθεί συζητήσει. Όσον αφορά τις εφαρμογές, δεν περιμένουμε το 2014-2020 για να απτυχθούν εφαρμογές. Ήδη στο έκτο πρόγραμμα πλαίσιο για, για την ε, έρευνα και την ανάπτυξη και στο επόμενο ε, προβλέπονται εργασίες για εφαρμογές στον τομέα των δρόμων, θαλασσίων μεταφορών ε, κινητής τηλεφωνίας, ε, ε, θαλασσίων μεταφορών, τραπεζικών συναλλαγών. Κάτι τελευταίο στο διεθνές επίπεδο. Ναι, έχουμε κάνει διαπραγματεύσεις, έχουμε στατική πρώτα απ' όλα μάλλον, όσον αφορά τις διάφορες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ενώσης. Έχουμε ήδη συμφωνία με Νορβηγία που συμμετέχει πλήρως στα προγράμματα. Σχεδόν έχουν τελειώσει διαπραγματεύσεις με την Ελβετία και έχουμε ήδη συμφωνίες συμβατότητας, παραδείγματος χάρη, με το Αμερικανικό σύστημα για να εξασφαλίσουμε τη συμβατότητα μεταξύ του GPS του Αμερικανικού και του Γαλιλαίου. Βλέπω ότι υπάρχουν πολλές πληροφορίες που πρέπει να σας δώσουμε, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να επανέλθουμε εδώ σε μία μήνυα ακρόαση για να σας δώσουμε ακόμα περισσότερες πληροφορίες. Ευχαριστώ, λέει Πρόεδρος. Ένα άλλο σύστημα για να ενημερώσουμε τις πληροφορίες μπορεί να είναι και εκείνο. Το λέω στον κύριο Φλαμάν. Να ετοιμάσετε ένα σημείωμα με απαντήσεις ακόμα αναλυτικότερες παρόλο που καλύψατε εκτενώς τις ερωτήσεις. Ε, ο κ. Μαρινέσκο δεν ξέρω αν έχει κάτι να προσθέσει. Παρακαλώ όμω πάρα πολύ σύντομα αν έχετε προσθέσει κάτι. Όχι, ευχαριστώ, λέει ο κ. Μαρινέσκο. Ευχαριστώ. Δεν θέλω να πω τίποτα τώρα. Δεν έχω τίποτα. Εκτό μικροφώνου, Πρόεδρο. 8 Μαου θα είναι έτοιμο αυτό το κείμενο. Λοιπόν, ευχαριστούμε όλου εκείνου που συμμετείχαν στην ανταλλαγή των απόψεων. Ήταν ενδιαφέρουσα συζήτηση. Επόμενο σημείο για το οποίο έχουμε μόλις ένα τέταρτο, σας παρακαλώ λοιπόν να περιοριστείτε ε, όσο γίνεται στις παρεμβάσεις σας. Αφορά το Δημιουργική Ευρώπη, το πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη, δίνουμε το λόγο στη Σίλβια Τικάου που είναι η συγγήτρια. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας τονίσω το πόσο σημαντικό είναι το να έχουμε ε, ε, τέτοιου είδου ε, ευκαιρίε ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων απασχόληση 4% το ΕΠ και 3,5% των, των θέσεων εργασία δημιουργούνται από τον τομέα του πολιτισμού. Τα ΜΜΕ πάντω έχουν ε, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν πρόβλημα για τους εξής λόγους. Υπάρχουν τα πνευματικά δικαιώματα. Επίσης υπάρχει και το πρόβλημα το ότι πολλές φορές ε, δεν είναι μαζικής παραγωγής τα πολιτικά προϊόντα. Οπότε ε, απουσιάζει και η εμπειρία ε, της θέσης τους σε εμπορία, λείπει η εμπειρία αναζήτησης χρηματοδότηση και πολλές φορές επομένως αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν υπάρχει αρκετή γνώση του αντικειμένου. Δεν έχουμε πάντως αρκετά στοιχεία σε σχέση με το γιατί οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν έχουν ε, αρκετή πρόσβαση στην δανειοδότηση. Έχουμε εδώ κάποιες προτάσεις για το πρόγραμμα. Και θα πρέπει επομένω να προσαρμοστούν και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην παγκοσμιοποίηση, στην ψηφιακή τεχνολογία και έτσι να δούμε τι θα γίνει με την πρόσβαση στα πολιτιστικά αγαθά πώς θα γίνει η αποθηκευσή τους σε ψηφιακή μορφή. Να δούμε ποια είναι η σχέση μεταξύ του τομέα των πολιστικών και του ιδιωτικού ε, τομέα, ούτως ώστε να βοηθηθεί η καινοτομία. Επίσης θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με συγκεκριμένους στόχους του προγράμματος, πώς θα βελτιωθεί η πρόσβαση των προσώπων με ειδικέ ανάγκες ε, στον τομέα τον, πολιτιστικό, τον δημιουργικό. Έχουμε εδώ δύο τροπολογίες, ούτως ώστε να ξεκαθαριστούν κάποια θέματα του προϋπολογισμού για τα εν λόγω προγράμματα. Επίσης, ε, έχουμε θίξει και το ζήτημα της συγχρηματοδότησης και όποιοι συμμετέχουν να μπορούν να προβούν στην αναγκαία προπαρασκευή για τους χρηματικούς και ανθρώπους πόρους. Ευχαριστώ την εισηγήτρια. Ο πρώτος που θέλει να πάρει το λόγο είναι ο συνάδελφος ο κ. Κέλλη. Εκτός μικροφώνου ο κ. Κέλλη. Micro, <laughs> I welcome the Creative Europe Programme proposal by the Commission. Πάρα πολύ θετική είναι η πρόταση της Επιτροπής. Η κυρίως αρμόδια Επιτροπή είναι η Επιτροπή των πολιτικών Θεμάτων που εκεί συμμετέχω και οπότε ε, βεβαίω έχουμε εδώ ε, κάποιε επιφυλάξει όσον αφορά το ποια είναι τα πλεονεκτήματα, ποια είναι τα μειονεκτήματα αυτού του προγράμματο. Μα θυμίζει το έρασμό αυτή η πρόταση, αυτό το πρόγραμμα. Πάντω, η αύξηση τη προκοδότησης είναι κάτι το θετικό. Έχουμε αυτή την 37%. Και έτσι αναγνωρίζεται στην πράξη η αξία της ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας. Οπότε τώρα έχουμε αυτή την ε, πολιτική πολυμορφία. Αυτό είναι ένα πλεονέκτημα. Αυτό μπορεί να μα οδηγήσει σε δημιουργία εκατοντάδων θέσεων εργασία. Εάν όμω προωθηθεί αυτή η υπόθεση με ε, σωστό τρόπο και όπω είπε και η συνάδελφο, έχουμε 5% του ΕΠ, 5% των θέσεων απασχόληση ε, που δεν καθόλου καταφρόνεται, δημιουργούνται από τον τομέα αυτό. Συμφωνώ με τόσο είπε η συγγήτρια, έχει δίκιο. Θα βελτιθεί το κείμενο εάν ε, πούμε ότι θέλουμε να καλύψουμε τις δημιουργικέ δυνατότητες των ε, αναπήρων. Επίσης, έχει δίκιο η συγκίτρια εκεί που λέει για την συνεργασία ιδιωτικού και δημόσιου τομέα και επίσης ε, η διαχείριση, η αποθήκευση του πολιτικού υλικού, όπως τα είπε. Όμως, να δούμε πώς θα υπάρχει συνέργεια με το Ευρωπαϊκό και δεν θα υπάρχει ε, παράλληλη χωριστή εξέλιξη. Έχουμε τέσσερις τροπολογίες. Καταθέσει για απλούστευση, θέσει απασχόλησης, πρόσβαση σε χρηματοδότηση, ιδίω όσον αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αθλητισμό, κοινωνικά, κοινωνικά μέσα και διεθνιστικό υλικό. Να σας πω δύο λέξει πάνω σε αυτά, γιατί είναι απλούστευση, τα έχουμε πει πολλέ φορέ εδώ στο Κοινοβούλιο και πρόσφατα ήρθαν και με βρήκαν ε, κάποιοι ψηφοφόροι μου και είπαν ότι δυστυχώ, δυστυχώς ε, πήγαν πάρα πολύ καλά γιατί όπως είναι τώρα η κατάσταση είναι αντιπαραγωγική και δεν τους βοήθησε κανένας. Θα πρέπει επομένω να δούμε πώ η διαδικασία, η διοικητική για τι ε, υποτροφίε για τα δάνεια θα βελτιωθεί. Με διάφορους τρόπους. Επίσης, όπως συζητήσαμε χθε για το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο, θα πρέπει να δούμε πώς θα καλυφθεί και αυτό το θέμα και πώς θα γίνει διαχωρισμός στην μεταχείριση και τη ρύθμιση των μικρών από τις μεσαίες επιχειρήσεις. Να έχουμε περισσότερους θύλακες, ε, κλάστερς και δεν πρόκειται να βοηθήσει μια βιομηχανία όταν δημιουργεί ευάλωτες θέσεις εργασίας. Ήδη σε κάποιες πόλεις όπως το Βαρκελόνη και το Βερολίνο και στον Κάλο στην Ιρλανδία έχουμε τέτοιους ε, θύλακες απασχόλησης. Γιατί χρηματοδότησε χρηματοδότηση τώρα οι, οι τραπεζές δεν εντονίζουν τώρα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δεν καταλαβαίνουν από πολιστικά και από δημιουργικά. Θα πρέπει η χρηματοδότηση να αμείβει τι πετυχημένες επιχειρήσει για τον αθλησμό τώρα να αναγνωριστεί σαν κομμάτι του πολιτιστικού τομέα και του δημιουργικού. Άρα θα πρέπει να αναφερθεί το YouTube και το Facebook και αυτά μπορούν να βοηθήσουν στο να προαχθεί ο τομέας των πολιτών, οπότε ελπίζουμε ότι και αυτά θα τα αναγνωρίσει το κείμενο. Τώρα τελευταίο και ίσως πολύ σημαντικό, αν θέλουμε να βοηθήσουμε τους, τα πολιτιστικά και τα δημιουργικά θα πρέπει να ξεκαθαριστεί ρητά ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα σύμβολα μνημονεύονται πάντως σε όλα τα προγράμματα. Γιατί πολλές φορές αναδύεται μόνο η εθνική πτυχή. Να, για παράδειγμα, Δευτέρα πρωί ερχόμουν εδώ και ένας υπουργός Ιρλανδός μου έλεγε για ένα πρόγραμμα ε, για τα σχολεία, το χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά πουθενά δεν αναφέρεται αυτό. Άρα, εδώ θα πρέπει να αλλάξει η κατάσταση και να βελτιωθεί. Σα ευχαριστώ κύριε Κέλεμ. Τακούλα και μετά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κουλά. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ο συνάδελφος Κέλλη έθεσε το ερώτημα αυτό εντελεχώς, δεν χρειάζεται πολλά να προσθέσω. Έχουμε πάρα πολλά καλά παραδείγματα για το συγκεκριμένο θέμα και το σχέδιο της κυρίας Τικάου αποτελεί άλλωστε ένα από τα σημεία προτεραιότητας της ε, θητείας μας, η προώθηση της ε, ψηφιακής ε, ατζέντα. Θα πρέπει λοιπόν αυτό να το κοιτάξουμε μέχρι το τέλος. Η δημιουργικότητα αυτή δεν προκύπτει από μόνη της, προκύπτει μόνο όταν υφίστανται οι απαραίτητοι όροι. Και ένας απαραίτητος όρος θεωρώ ότι είναι και η ψηφιακή ενιαία αγορά. Το ερώτημα λοιπόν θα πρέπει να επιληθεί κατά αυτόν τον τρόπο το αυτό. Σήμερα υπάρχουν διαφορετικά συστήματα στα διάφορα κράτη και αυτό θα πρέπει να απλοποιηθεί ως διαδικασία προκειμένου να υπάρχει καλύτερη ορατότητα. Επίσης, πολύ σημαντικό είναι να δημιουργηθεί μια στενή σύνδεση με τη Στρατηγική Ευρώπη 2020 και κατά την παρακολούθηση των προγραμμάτων αυτών θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να διαπιστώσουμε ότι δημιουργείται ένα μεγάλο πλαίσιο. Με τον τρόπο αυτό λοιπόν θα πρέπει να δημιουργηθεί προστιθέμενη αξία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επίσης πολύ σημαντικό είναι το εξής. Στο σχέδιο αυτό γίνεται σαφής αναφορά στην πολυγλωσία και στην πολιτισμική ποικιλία και στην ε, συμμετοχή συγκεκριμένων ομάδων, όπως για παράδειγμα η ανάπηροι. Οι ψηφιακές υπηρεσίες σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να αυξηθούν και σίγουρα θα αυξηθούν και αυτό ασφαλώς και θα αποβεί προς όφελος όλων των κοινωνικών ομάδων και όλων των Ευρωπαίων πολιτών. Ιδιαίτερα το θέμα της προσβασιμότητας είναι πάρα πολύ σημαντικό και ολοκληρώνω, Πρόεδρε, Υπάρχει λοιπόν αυτή η επισκόπηση. Καθοριστική σημασία είναι η Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Ενιαία Αγορά. Θα πρέπει τα ευρωπαϊκά κράτη να συμφωνήσουν επί μια καλύτερης συνεργασία προκειμένου να αποφεληθεί και η ευρωπαϊκή ανάπτυξη. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Σίλβερ εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει το λόγο, αλλά παρακαλώ συνοπτικότατη, διότι θα πρέπει να ξεκινήσει λίγα λεπτά η ψηφοφορία. Thank you. Σας ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να μιλήσω. Θα είμαι, το συντομότερο, θα είμαι όσο δυνατόν συντομότερη. Θα ήθελα καταρχάς να διευκρινίσω ότι καλωσορίζουμε τις γνωμοδοτήσεις του Κοινοβουλίου και ότι συμφωνούμε με πολλές από τις προσεγγίσεις. Να περιοριστώ ίσως σε κάποια μικρά σχόλια για όσα ήδη αναφέρθηκαν. Ιδιαίτερα για θέματα απλούστευσης, μιας και ξεκινήσαμε ήδη μια σημαντική διαδικασία απλούστευσης ε, με τις ηλεκτρονικές ε, με τα ηλεκτρονικά έντυπα και θέλουμε να το συνεχίσουμε εδώ με τα καταποκοπή ποσά σε ό,τι αφορά τη διευκόλυνση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και του δημιουργικού κλάδου προκειμένου να μην ε, ωφεληθούν μόνο οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αλλά και οι πολύ πολύ μικρές επιχειρήσεις και αντιλαμβανόμαστε πολύ καλά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις αυτές σε ό,τι αφορά την υποβολή αιτήσεων για χρηματοδοτήσεις ε, από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήδη σε ό,τι αφορά θέσει εργασία, προωθούμε τη λειτουργία, την δημιουργία κλάστερ και συμπράξεων ε, δημοσίου και δυτικού τομέα και αυτό είναι κάτι το οποίο θα το συνεχίσουμε στο μέλλον. Σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στη χρηματοδότηση τώρα, θα ήθελα να τονίσω τα μοναδικά χαρακτηριστικά της ε, του μέσου διευκόλυνσης εγγυήσεων που σκοπό έχει να αλλάξει την νοοτροπία του τραπεζικού κλάδου έναντι των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στον κλάδο τον πολιτισμικό και τον δημιουργικό προκειμένου να αποφευθεί μία κατάσταση όπου θα πρέπει να βάζουν προσωπικά εγγυήσει για να λάβουν δάνεια τέλος σε ό,τι αφορά τη χρήση των κοινωνικών ε, media και του αθλητισμού θα υπάρχει έντονη σύνδεση μεταξύ του Erasmus for All που και του Creative Europe σε ό,τι αφορά τα ζητήματα που ε, τέθησαν για τα σύμβολα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε και ενέκρινε πρόσφατα μία νέα τέτοια ταυτότητα, αλλά θα χρησιμοποιήσουμε την ετικέτα ε, που χρησιμοποιείται εδώ και 20 χρόνια μέχρι τα τέλη του 2013. Και ένα τελευταίο σημείο. Το πρόγραμμα αυτό όντως συγκαταλέγεται στο πρόγραμμα Ευρώπη 2020 και δεδομένων και των ε, πολλών θέσεων εργασία υψηλή εξειδίκευση ε, στον κλάδο αυτό, είναι κάτι που θα πρέπει να υποφεληθεί από την ψηφιοποίηση και την παγκοσμιοποίηση και ασφαλώ θα πρέπει να λάβει την υποστήριξή μα προκειμένου να μπορέσει όντω να αντράξει τι ευκαιρίε αυτέ που ανοίγονται. Ευχαριστώ. Eh, Σα ευχαριστώ, συνάδελφο δεν θέλει να παρέμβει, προσπαθεί να βοηθήσει την Προεδρία στην ξενονόηση του χρόνου. Προθεσμένη υποβολή τροπολογιών είναι 3 Απριλίου. 3 Απριλίου στι 12 το μεσημέρι. Πριν ολοκληρώσουμε αυτό το κομμάτι των εργασιών μα, συνεχίζοντα μια παράδοση που ο πρόεδρο Ρόιλ είχε ξεκινήσει, θέλουμε ευχηθούμε και εμείς χρόνια πολλά, στον συνάδελφο Ματσικίεβιτς, που έχετε γενέθλια σήμερα. Συγχαρητήρια και χρόνια πολλά σε εσά, κύριε interrompere. Μπορούμε να διακόψουμε. Ένα μικρό διάλειμμα για να πάρει ο καθένας ε, τον κατάλογο συμφοριών. Ε, Ας ετοιμαστούμε λοιπόν για τις ψηφοφορίες. Ας κάνουμε πρώτα μία δοκιμή, να δούμε αν λειτουργεί το μηχάνημα. Παρακαλώ να ψηφίσουμε τώρα δοκιμαστικά. Ας κάνουμε προσωμείωση ψηφοφορίες, αν συμφωνείτε. Ας ψηφίσουμε Ποιος είναι υπέρ. Κατά, αποχές. La votazione chiusa. Πέρας. Φαίνεται ότι δουλεύει. Δεν ξέρω τι δοκιμάσαμε, αλλά ό,τι δοκιμάσαμε δούλεψε. Πρώτη ψηφοφορία υπάρχει κάποιο διαδικαστικό. Και ως Πετικόβα ήθελα να σας πω, κυρία Πρόεδρε, δεν μπορώ να ψηφίσω, δεν έχω την κάρτα μου, θα εξακολουθώ, θα ψηφίσω. Λοιπόν, αν μπορείτε να μετρήσετε την ψήφο μου, γιατί ε, δεν έχω την κάρτα μαζί. Υπάρχει χορός ε, αποδοκιμασίας, λέει Πρόεδρος, Πρόεδρος, παρόλα αυτά θα συνεχίσουμε. Πρώτα ξεκινάμε από την εισηγήτρια την κυρία Τσικάου αγορά ψηφιακής ανταγωνιστικότητας. Ξεκινάμε τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 4. Υπέρ. κατά αποχές εγκρίνεται 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 1 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 11 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 15 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 17 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 5 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 19 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 21 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 22 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 25 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 31 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 33 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 34 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 35 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 36 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 37 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Τροπολογία 38 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 39, προφορική τροπολογία, τσουκάλι. Συνάδελφοι, μπορείτε να προτείνετε προφορική τροπολογία. Αυτό που προτείνω, μία προσθήκη να προσθέσουμε το εξή στην Αντροπολογία 39. Υπενθυμίζει την ουσιαστική δέσμευση μείωση των ψηφιακών κενών αναφευρισμού ψηφιακού και τομένων κενών αρμοδιοτήτων κατά το ίμιση μέχρι το 2015. Ας ψηφίσουμε λοιπόν τροπολογία 39 με την προφορική τροπολογία. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται, συμβαστική 6 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 42 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 43 τροπολογία 43 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 44 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Τροπολογία 46 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 47 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 48 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 49 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 50 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 52 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 53 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 29 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Μκο 23 έλεγχος μκο 16 ηλεκτρονικός έλεγχος υπέρ λέει η πρόεδρος άρχεται η ψηφοφορία La votazione chiusa. Πέρας. Εγκρίνεται. Με μικρή διαφορά, αλλά εγκρίνεται. ΕΜΚΟ 23 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται πολιτισμού 2, κουλτ 2 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, κουλτ 4 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, κουλτ 6 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, κουλτ 17 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, κουλτ 7 υπέρ, Α, έκανα λάθο. Κουλτ 8, υπέρ. Κατά. Αποχέ, εγκρίνεται. Κουλτ 9, υπέρ. Κατά. Αποχέ, εγκρίνεται. Κουλτ 10, υπέρ. Κατά. Αποχέ, εγκρίνεται. Κουλτ 11, υπέρ. Κατά. Αποχέ, εγκρίνεται. Τζούρι 1, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται τζούρι 2 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τζούρι 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τζούρι 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικός άρχεται ψηφοφορία ηλεκτρονική ψηφοφορία πέρας Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται. Νομίζω ότι η συγγήτρια αξίζει με συγχαρητηρίων, πολλών συγχαρητηρίων. Για αυτή την ψηφοφορία, την ομοφωνή, ζήτησε, ζήτησε το λόγο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους, ιδιαίτερα τους κοιότες εισηγητές και τη γραμματεία για όλη την καλή δουλειά του. Ε, Μπουτικόφερ. Κύριε Μπουτικόφερ, ζητήσατε το λόγο, όχι. Εκτό μικροφώνου και Μπουτικόφερ, οι διερμηνεί δεν τον ακούν. E Σα ευχαριστώ όλου. Τελειώσαμε το πρώτο απλούστατο σημείο, μετά έχουμε τα επόμενα. passiamo al voto del rapporto Crossman. Έκθεση Κόσμαν. Τροπολογία 1 υπέρ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 1 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 4 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 9 με προφορική τροπολογία που διαβάσατε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 11 υπέρ κατά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 κατά αποχές νομίζω ότι απορρίπτεται συμβαστική 36 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 6 λιπρόδρος υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 45 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 46 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 47 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 48 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 49 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 51 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 52 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 53 σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ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 Συμβαστική 8 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 64 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 9 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 66 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 67 με προφορική τροπολογία που έχετε στο κείμενο υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε όλο το κείμενο. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας εγκρίνεται. Passiamo al Λάγκεν. Πάμε στο επόμενο. Τροπολογία 41 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 5 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 42 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 6 υπέρ. Με προφορική τροπολογία η 6 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 7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 21. Έλεγχος. Άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ηλεκτρονικός έλεγχο για την 21. Πέρα. Υπέρ 20 κατά 30. Ναι, μάλιστα. Απορρίπτεται. 22 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 23 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 25 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 24 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 26 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 1 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Έλεγχος όσον αφορά την 1. Πέρας 36 υπέρ, 15 κατά εγκρίνεται. 28 υπέρ. Κατά. 28. 28. 28 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος για την 28. 37 υπέρ, 18 κατά. Ένα σελκ παραπάνω, δεν αρέσει τίποτα. Εγκρίνεται. 29 υπέρ, κατά. Αποχές απορρίπτεται. 2 υπέρ, κατά. Απορρίπτεται. 30. Έλεγχος για τη 2. Votazione aperta. Πέρας. 30 υπέρ, 25 κατά. Εγκρίνεται. 3. Σε δύο ξεχωριστά τμήματα. Πρώτο τμήμα της υπέρ. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 31 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 33 α συγγνώμη 4 4 πηδήξαμε το 4 υπέρ σε τρία τμήματα 4 σε τρία τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές συγκρίνεται. δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές φαίνεται να απορρίπτεται θα κάνουμε έλεγχο δεύτερο τμήμα του 4 ηλεκτρονικός έλεγχος πέρας ψηφοφορίας 30-23 τρίτο τμήμα υπέρ κατά Αποχές εγκρίνεται. 35. 35 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 36 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 37 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 38 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 39 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία, ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. 54 ψήφοι υπέρ και μία αποχή. Ομόφωνα. Συγχαρητήρια. quest Καλώς ολοκληρώθηκε η ψηφοφορία. Σας ευχαριστώ όλους, εισηγητές και ψηφοφόρους. Πάμε στην έκθεση για εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, εισηγήτρια. Ο Τάκης Χατζηγεωργίου είναι ο εισηγητής δεν είναι εδώ ο εισηγητής ο κ. Χατζηγεωργίου δεν είναι εδώ Α, είναι εδώ Τέλεια Ο εισηγητής λοιπόν έχει το λόγο Λοιπόν, εμείς ε, θεωρούμε ότι πρέπει να υποστηριχθεί αυτό το κείμενο της Επιτροπής για καλύτερη διαχείριση του υφιστάμενου μηχανισμού παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και αυτό γιατί πιστεύουμε ότι <coughs> ε, Περιμένετε μισό λεπτό παρακαλώ για να διάσει η αίθουσα. Όσοι είναι να φύγουν την αίθουσα να φύγουν. Bene. Καλώς. μπορούμε να ξεκινήσουμε. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Έλεγα λοιπόν ότι εμείς υποστηρίζουμε <clears throat> την πρόταση της Επιτροπής για καλύτερη διαχείριση του υφιστάμενου μηχανισμού παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου γιατί βρίσκομαι πως είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Θεωρούμε ότι ενισχύει τις προσπάθειες για συντήρηση ε, του κλίματος στον πλανήτη μέσα στα πλαίσια τα οποία όλοι αναζητούμε. Θεωρούμε ότι ενισχύει τις προσπάθειες των κρατών για να κρατήσουν τα επίπεδα των ρήπων ε, στο σημείο εκείνο που είναι επιτρεπτό υπό τις συνθήκες και εκτιμώντας απλώς ότι κάποια σημεία στην πρόταση μπορούν να χρειαστούν περαιτέρω προβληματισμό θέλουμε να καταθέσουμε κάποιες απόψεις. Το πρώτο που θέλουμε να πούμε είναι ότι στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου πρέπει να αποφευθεί οποιαδήποτε περαιτέρω επιβάρυνση κατά αυτή την περίοδο των κρατών μελών ένα και της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. Να υπάρξει μια έκφραση ε, ανησυχίας, έγνοιας γύρω από αυτό το σημείο σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Επιπλέον θα πρέπει να μας προβληματίσει το γεγονός ότι ακόμα να τεθεί σε ισχύ η δέσμευση για δημιουργία του Πράσινου Ταμείου που στοχεύει στην ενίσχυση των προσπαθειών των φτωχών χωρών για καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών. Θέλουμε επίσης να επισημάνουμε ότι είναι καλό να προβληματιστούμε για την καταλληλότητα ή και βιωσιμότητα του Ευρωπαϊκού Συστήματος Εμπορίας Ρήπων, που η αρχική του φιλοσοφία η οποία λέει ότι ο ρηπαίνων πληρώνει, θα πρέπει να έχουμε μια αυξημένη έγνοια μην μετατραπεί αυτό κάποια στιγμή αντί ο ρηπαίνων πληρώνει να γίνει ο πληρώνων ρηπαίνει. Γιατί ασφαλώς δεν είναι αυτό στόχος κανενός. Τέλος θέλω να επισημάνω ότι η πρόταση δεν λαμβάνει υπόψη το γεγονό ότι η Κύπρος και η Μάλτα έχουν ήδη ενταχθεί στο παράρτημα 1 του πρωτοκόλλου του Κιώτο και η σύσταση της Επιτροπής φαίνεται ότι γράφτηκε πριν να συνυπογράψει η Κύπρος και η Μάλτα το συγκεκριμένο πρωτόκολλο. Κλείνω επαναλαμβάνοντας ότι θα επανέλθουμε ίσως αφού ακούσουμε και τους ε, εισηγητές σήμερα εδώ σε επόμενη συνεδρία για να δούμε πώς γινόμαστε πιο πρακτικοί στην υποστήριξη της μεγάλης προσπάθειας που καταβάλλεται να κρατηθούν οι ρήποι στα κράτη-μέλη και όχι μόνο ε, στο βαθμό που μπορεί να είναι επιτρεπτό και ανοιχτό σήμερα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Όλ έχει ζητήσει το λόγο. Έχετε το λόγο. Thank you, Madam President. Um... Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλωσορίζω ιδιαίτερα τον κανονισμό αυτό, γιατί είναι κρίσιμο να γνωρίζουμε κατά πόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη ακολουθούν τους στόχους που έχουν τεθεί για την απεξάρτηση από τον άνθρακα και επίσης επειδή ζητά από τα κράτη-μέλη να παρέχουν διαφανείς πληροφορίες για τον τύπο και το ποσό υποστήριξης που παρέχεται στις αναπτυσσόμενες χώρες και αυτό είναι πραγματικά κλειδί για να αυξηθεί η αξιοπιστία της Ένωσης στις χώρες αυτές και για να αξιολογηθεί κατά πόσον τηρεί τις δεσμεύσεις της η Ένωση Υπάρχουν ωστόσο κάποιοι τομεί όπου θεωρώ ότι θα μπορούσαμε να ενισχύσουμε τον κανονισμό. Καταρχά. είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει μακροπρόθεσμη προοπτική και να δούμε κατά πόσο η Ένωση και τα κρατημέλη ε, ακολουθούν την πορεία τους για να ε, ανταποκριθούν στους στόχους του μακροπρόθεσμου του 80-95% μέχρι το 2050. Ψηφίσαμε και την προηγούμενη εβδομάδα μία πορεία μέχρι το 2050 σε ό,τι αφορά τους στόχους για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου σε ό,τι αφορά το 60% το 2040 και τα λοιπά σε σχέση με τα επίπεδα του 90. Νομίζω ότι καλό θα ήταν ο κανονισμός να ζητά από τα κρατημέλη να παρακολουθούν και να αναφέρουν πώς εξελίσσονται οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και κατά πόσον πληρούν τους όρους που έχουν τεθεί και τους στόχους της Ένωσης. Ιτάλος υφίσταται ο κίνδυνο, να τρέχουμε τελευταία στιγμή και να είναι πάρα πολύ δύσκολη η εφαρμογή και πολύ δαπανηρή. Κατά δεύτερον, η πλήρης ε, κατάργηση των αερίων του θερμοκηπίου θα σημαίνει ότι θα πρέπει να δραστηριοποιηθούμε από το σύστημα ETS και θα πρέπει να δούμε τι γίνεται και στον τομέα που δεν εντάσσεται στο ETS για τη γεωργία, δεν αναφέρεται τίποτα για τα κτίρια που ε, εκπέμπουν το 40% των ε, εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Γι' αυτό λοιπόν καλό θα ήταν να συμπεριληφθεί στον κανονισμό η υποχρέωση για τα κράτη-μέλη να αναφέρουν τι γίνεται λοιπόν για την εξοικονόμηση ενέργεια στα κτίρια, τι γίνεται με τι ανανεώσιμε πηγέ. Αυτές οι πληροφορίε υπάρχουν, δεν του ζητούμε να τις συλλέξουν επιπλέον, γιατί υποβάλλουν τις σχετικές αναφορές σε άλλο επίπεδο. Καλό θα ήταν λοιπόν να τις υποβάλλουν και στο πλαίσιο αυτό. Δεν θα σημαίνει επιπλέον φόρτο εργασίας, γιατί έτσι και αλλιώς τις υποβάλλουν. Τέλος το συνέδριο στο Κανκούν το 2010 τα μέλη συμφώνησαν τα συμβαλόμενα μέλη να υποβάλουν αναφορές για την υποστήριξη που παρέχουν προς ε, τις αναπτυσσόμενες χώρες. Οι πληροφορίες αυτές αποφασίστηκε ότι θα πρέπει να είναι το δυνατόν πιο διαφανής. Θα θέλαμε λοιπόν και εδώ να αναφέρεται ότι αυτή η οικονομική και τεχνολογική αρρωγή είναι πρόσθετη στα συνηθισμένα μέτρα και πραγματικά συνεισφέρει στην τεχνογνωσία στις αναπτυσσόμενες χώρες, αλλά και στην περιβαλλοντική και κοινωνική ε, ακαιρεότητά τους. Άρα, λοιπόν, θα μπορούσε να προβλέπετε καλύτερη υποχρέωση αναφορών στον κανονισμό σε ό,τι αφορά το τι κάνει η Ένωση και τα κράτη-μέλη προ τι αναπτυσσόμενε χώρες σε σχέση με αυτά που έχουν συμφωνηθεί και στο Κανκούν. Ευχαριστώ κυρία Τζόρνταν. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Πολλά από τα έγγραφα τα οποία έχουμε εδώ μιλούν για την αλλαγή του κλίματος και σε σχέση με τον χάρτη πορείας 2050 μιλάμε για κάποια βασικά στοιχεία γιατί δεν μπόρεσα να διαβάσω όλο το Έγραφα Να σα πω τι θέσει του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματο. Πρόκειται για ένα έγγραφο το οποίο αφορά κυρίω την Επιτροπή Περιβάλλοντο. Αλλά εμεί θα πρέπει να δούμε εκείνα τα θέματα τα οποία αφορούν τη δική μα Επιτροπή, τι δικέ μα αρμοδιότητε. Διότι συμφωνώ 100% με αυτό το οποίο ανέφεραν οι προλελήσαντε συνάδελφοι. Όμω α προχωρήσουμε με προσοχή και α επικεντρώσουμε την προσοχή μα στα θέματα δική μα αρμοδιότητα. Όλοι αυτό το οποίο θέλουμε είναι το σύστημα να είναι αποτελεσματικό και απλό. Και επίση, ε, από όσο μπορούσα να διαβάσω, θεώρησα ότι είναι πάρα πολύ πολύπλοκη αυτή η πρόταση και το πιο σωστό είναι να κάτσουμε με τους ε, σκιώδεις ηχητές και να κοιτάξουμε τι θα γίνει με την, ε, με την απλούστευση. Ε, θα πρέπει με τη συνάδελφο να κάτσουμε και να κωδικοποιήσουμε, να αναβάλουμε σε, ένα εγγραφό όλα τα, τα, τα, τα στοιχεία και θα πρέπει να περικόψουμε τις διάφορες διοικητικές διαδικασίες. Εδώ πάντως ε, αναφέρεται το ότι η βιομηχανία δεν θα πρέπει να επιβαρύνεται με, με, με τέτοιες τυπικότητες, αλλά έτσι κι αλλιώς οι διοικητικές υπηρεσίες ε, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι γίνονται περικοπές, η ρίγνωση του, του, του, του δημόσιου τομέα. Οπότε γι' αυτό το λόγο δεν θα πρέπει να επιβαρύνουμε περισσότερο ούτε την βιομηχανία, ούτε τους επιχειρηματίες, αλλά ούτε και την διοίκηση. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ εύστοιχο το ότι εδώ πέρα μιλούμε για την εμπορία εκπομπών. Θα πρέπει επομένως αυτό το σύστημα να το αξιοποιήσουμε. θα πρέπει να δούμε ε, πώς θα αξιοποιήσουμε τους, ε, τους πόρους που υπάρχουν κάτι άλλο τώρα στο έγγραφο επίσης αναφέρεται η προετοιμασία κάποιων προγραμμάτων για την μείωση των εκπομπών του διοξιδίου. Στόχος είναι να γίνει αυτό πριν το 2050. Το Κοινοβούλιο το συζήτησε την περασμένη εβδομάδα και αναφέρθηκε ότι η σχετική στόχοι δεν είναι δεσμευτική Αυτό να διατυπωθεί στο νομοθετικό έγγραφο. Να μην είναι αυτή η στόχη δεσμευτική, αυτή η στόχη του 2050. Κάτι άλλο τώρα. Θα ήθελα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας ενημερώσει παραπάνω όσον αφορά την σύγκριση του συστήματος που ισχύει σε εμά με αυτό που ισχύει στις πολιτείες. Ευχαριστώ. Η Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ. Ο Κλοντ Τούρμς έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. I, Νομίζω ότι τα σημεία που ανέφεραν οι συνάδελφοι σε σχέση με την υποβολή αναφορών και για την συγκέντρωσή τους προκειμένου να μην έχουμε δέκα μικρές εκθέσεις αλλά μία συνεκτική έκθεση αναφορά. Αυτό θα συνεπάγεται όχι μόνο λιγότερο γραφειοκρατικό άχθος αλλά και πολιτικός πώς είναι πιο σωστό αυτό γιατί σε μία στιγμή αποκρισταλώνεται η όλη εξέλιξη. Άρα είμαι σαφώς υπέρ της πρότασης αυτής συμπεριλαμβανομένου του στοχου 2020 20 και τα ποσοστά ανανεώσιμων θα βοηθούσαν προς την κατεύθυνση αυτή. Φυσικά έχουμε και το θέμα του Κανκούν και της κλιματικής στρατηγικής και κατά πόσο εντάσσεται αυτό μακροπρόθεσμα στον οδικό χάρτη για το 2050. Νομίζω ότι και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό είναι το θέμα των εκπομπών του ναυτιλιακού κλάδου, γιατί αυτό θεωρώ ότι αποτελεί την επόμενη μεγάλη διεθνή μάχη Ξέρετε ότι ο ναυτιλιακός κλάδος δεν καλύπτεται από καμία νομοθεσία για το κλίμα σήμερα και είναι πραγματικά πολύ αναποτελεσματικός ο τρόπος καύσεως πετρελαίου. Θα πρέπει να δοθεί λοιπόν ένα σαφές μήνυμα προς την ναυτιλία. Αυτά τα τέσσερα σημεία ήθελα να αναφέρω. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ο συνάδελφος Σκέλη. Α, συγγνώμη. Ο κ. Πρόντι πρώτα. Ευχαριστώ Πρόεδρε να υπογραμμίσω ιδιαίτερος το GMES ε, τι δυνατότητες έχει για τον υπολογισμό των εκπομπών για τη μέτρηση των εκπομπών. Ο δορυφόρος δύναται να δείξει τη συγκεντρώση στην ατμόσφαιρα των αερίων του θερμοκηπίου και μπορεί τι το τρόπος να βοηθήσει να ε, δείξει, να μας οδηγήσει σε πλήρη καταγραφή των εκπομπών, σαφή εικόνα και σε πραγματικό χρόνο να μπορούμε να μετρήσουμε τις εκπομπές και κάθε χώρας. Και αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και να παρακολουθηθεί διότι μπορεί να μας δώσει πολύ λεπτομερή ε, και ακριβή στοιχεία. Ως παρατηρήση θέλω να πω ότι η τομεκή των εκπομπών που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν επιτρέπει να είμαστε τόσο ακριβείς και τόσο έγκαιρα να σημειώνουμε τις εκπομπές. γενικότερη πειθαρχία θα μπορούσε να παρακολουθηθεί ευκολότερα. Εξηγούμε. Αν κάθε ένας που χρησιμοποιεί ορυκτά κάψιμα υποχρεούται να έχει σχετικές άδειες εκπομπών, τότε όλα θα προχωρούσαν πολύ πιο, αργά, πολύ γρήγορα συγγνώμη, και θα ήταν όλη η κατάσταση πολύ απλούστερη όλη η παρακολούθηση πολύ απλούστερη. Ο συνάδελφος Κέλλη έχει το λόγο τώρα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Εν συντομία. Ένα σημείο ήθελα να θίξω. Ο εισηγητής αναφέρθηκε στο ότι θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, να μην ε, κινούμαστε από μία ε, κατεύθυνση όπου πληρώνει ο ρηπαίνο στο ότι πληρώνει τελικά ο Αυτό να το προσέξουμε γιατί προφανώ δεν έχει νόημα να γίνει κάτι τέτοιο να επαναλάβω το σημείο που αναφέρθηκε ότι θα πρέπει να υπάρξει ε, καλή καταγραφή, καλή υποβολή αναφαρών, δημοσίευση των στατιστικών στοιχείων ανά κράτος μέλος, προκειμένου να υπάρχει μια ενδιάμεση παρακολούθηση μεταξύ της τωρινής στιγμής και του 2050 και θα Ήθελα να τονίσω και αυτά που αναφέρθηκαν για τα κτίρια, 40% οι εκπομπές, η κατανάλωση. Και επίσης ε, να τονίσω αυτό που είπε ο κύριος Τούρκμες για την αυτιλία. Αυτά λοιπόν θα πρέπει όλα να συμπεριληφθούν αν θέλουμε να πετύχουμε τους συνολικούς μας στόχους μέχρι το 2050. Σας ευχαριστώ, συνάδελφε Κέλλη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να πάρει το λόγο εκπροσωπός της. Uh, ναι, κυρία Πρόεδρε, αυτό που θα ήθελα να σας τονίσω είναι ότι όταν μιλούμε για ολιστική προσέγγιση, εννοούμε να υπάρχει μία και μόνη πρόταση κανονισμού και να ισχύουν όλα όσα ήδη προβλέπονται για τον μηχανισμό υποπτίας και παρακολούθησης και επίσης να ισχύει ό,τι ήδη έχει θεσπιστεί διεθνώς για τις δεσμεύσεις διεθνώς και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά το, τη δέσμη μέτρων για το κλίμα, ό,τι, ό,τι έχει προσθεθεί επομένως τώρα για ό,τι, ό,τι έχει προσθέσει αυτό που υπήρχαν. Αυτό εννοούσαμε τώρα για να επανέλθουμε στο θέμα των επιπτώσεων. Εμείς με αυτή την πρόταση κάναμε και μία είναι εντελεχή έκθεση επιπτώσεων και είπαμε ότι απευθύνουμε αυτό ότι, ότι, ότι δεν υπάρχει άμεση επίπτωση σε ε, ΜΜΕ και στην βιομηχανία αλλά στα κράτη, η επιπτώση είναι για τα κράτη-μέλη επί τη βάση της υπάρχουσας συλλογής στοιχείων. Επομένως, για αναφορές, εκθέσεις, εποπτεία. Λάβουμε υπόψη το τι ήδη ισχύει. Και επομένω θα είναι πολύ περιορισμένη η επιβάρυνση των κρατών μελών. Δεν έχουμε άμεσε επιπτώσει από αυτόν τον κανονισμό για ΜΜΕ και βιομηχανική Και για τα κράτη-μέλη είπαμε ότι πάμε στο 3,5, στα 3,5 εκατομμύρια για τα 27 κράτη-μέλη. Αυτό είναι βέβαια ένας μέσος όρο. Αλλά σε σχέση με αυτό το οποίο θέλουμε να πετύχουμε, όλοι έχουμε αυτό το στόχο. Και έτσι θα πετύχουμε να μειωθούν οι εκπομπές σε σχέση με το στόχο του 2020 αλλά και με στόχο με ορόσημο του 2050 όμως χρειάζονται κάποιες ελάχιστες επενδύσεις για να κάνουμε τις μικρές προσαρμογές που χρειάζονται στην δράση των κρατών μελών για αναφορές και υποπτία. Τώρα όσον αφορά το Green Fund ξέρουμε τι αποφάσεις έχουν ληφθεί. Προχωρούμε ταχαίως στη συγκρότηση αυτού του ταμείου και οι προσδοκίες παραμένουν σημαντικές. Τώρα όσον αφορά τις θαλάσσιες μεταφορές είπαμε ότι γίνονται προσπάθειες σε κάθε επίπεδο και μόλις υπάρξει κάποιο κείμενο που θα μπορέσουμε να καθορίσουμε τις προϋποθέσεις της ε, εποπτείας θα προχωρήσουμε όσο πιο ωραία γίνεται. Για τα κτίρια τώρα ήδη τηρήσαμε τη διεθνή μας δέσμευση για την υποβολή των εκθέσεων, των αναφορών. Θα κάλυψε επομένως ήδη ο κανονισμός. Τώρα όσον αφορά τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης, όπως θα το έχετε ήδη διαβάσει στην έκθεση πρόοδου του Οκτωβρίου 2011 ξέρετε ότι υπάρχει κίνδυνος να υπάρχουν τέτοιες επιπτώσεις όμως εμείς θεωρούμε ότι θα ελέγξουμε αυτές τις επιπτώσεις εκθέσεις για εποπτεία και θα υπάρξουν και κάποιες πολιτικές, κάποια μέτρα που θα ληφθούν. Και έτσι, με τα υπάρχοντα μέτρα ή και με κάποια παραπάνω, θα μπορέσουμε να πετύχουμε το στόχο μας. Για το GMS, για το GMS, GMS προσπαθούμε να συγκροτήσουμε μια τέτοια υπηρεσία για την κλιματική αλλαγή. Και μελετούμε ποια είναι τα πλεονεκτήματα μιας τέτοιας κίνησης. Και η εμπειρία μας από την υπάρχουσα υπηρεσία κατατείνει στο ίδιο συμπέρασμα ότι θα υπάρξουν πλεονεκτήματα. Τώρα, για τον κύριο Χατζηγεωργίου, ε, σε σχέση με Κύπρο και Μάλτα, σε σχέση με όσα μα είπε, ναι, γνωρίζουμε ότι έχουμε το COP15 και COP17. Σημαίνει ότι θα πάμε για ε, να διέπει Μάλτα και Κύπρο το καθεστώς ε, του στόχου 1 του παραδείγματος 1 και επομένως δεν νομίζω θα υπάρξει κάποιο πρόβλημα που να μας απασχολεί και να σας απασχολεί τώρα όσον αφορά το ότι θα πρέπει να έχουμε κάποια μακρόπνευμα προοπτική στο κείμενο γίνεται παραπομπή στο χάρτη πορείας για το 2050 το θέμα συζητείται τώρα στο Συμβούλιο αλλά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τον κανονισμό λαμβάνει υπόψη την αύξηση της ε, θερμοκρασίας κατά δύο βαθμούς και είπαμε ότι ναι, η στόχη αυτή δεν είναι δεσμευτική, αλλά στην πράξη πρέπει να τηρηθούν τα σχετικά μέτρα για να μπορέσουμε να πετύχουμε τον κοινό μας στόχο. όλα όσα σήμερα αναφέρονται συμπληρώνουν. Είναι στο μήκο κύματο των όσων και εμεί θέλουμε να κάνουμε. Αν έχετε κάποιε συγκεκριμένε ε, ερωτήσει, ευχαριστώ να απαντήσω. Ευχαριστώ. Ο Χατζηγεωργίου έχει το λόγο για να δώσει απαντήσει. Ε, υπόψη τα όσα ελέγχθησαν που δείχνουν ότι είμαστε όλοι προς ε, κοινό στόχο, ανεξάρτητα από επιμέρους ε, προσθέσεις ιδεών. Ε, θεωρώ ότι απλώς εντάχει πρέπει να υπογραμμίσω όσα έχω σημειώσει και που βρίσκω και εγώ ότι πρέπει να μας απασχολήσουν θετικά, που είναι η αναφορά στις εκπομπές ρήπων από κτίρια από τη Γεωργία και από την Ναυτιλία, Άκουσα με ενδιαφέρον την σκέψη να κάνουμε σύγκριση μεταξύ του δικού μας συστήματος και του συστήματος των Ηνωμένων Πολιτειών. Θα λάβουμε υπόψη την ε, αναφορά για τις βιομηχανίες που χρησιμοποιούν οριχτά καύσιμα και νομίζω ότι η μόνη ε, διαφορά άποψη που μπορεί να έχω είναι στην τοποθέτηση που έχει γίνει να μην είναι δεσμευτική η στόχη ε, του 2050. Τίποτα βέβαια δεν μπορεί να είναι ε, θέσφατο, όμως θεωρώ πως οι δεσμεύσεις έχουν την σημασία τους. Επιφυλασσόμαστε για την επόμενη συνεδρία να έρθουμε έχοντας κατά νου και τις προτάσεις που έχουν ακουστεί σήμερα εδώ. Ευχαριστώ. Καλώς. Ολοκληρώθηκε η συζήτησή μας. Το σχέδιο γνωμοδότησης δεν είναι ακόμα διαθέσιμο, αλλά έχουμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχουμε το σχέδιο εκθέσεως επίσης που είναι διαθέσιμα. Η ημερομηνία για τις τροπολογίες 5η 12 Απριλίου, 12 το μεσημέρι. Πάμε στο επόμενο, στην επόμενη έκθεση. Ο συνάδελφος Σιμάσκι δεν είναι εδώ. Ο συνάδελφος Τσίτσεστερ θα μιλήσει εν ονόματι του. Ευχαριστώ Πρόεδρε και κύριε Σιμάνσκι. Ζητά συγγνώμη που δεν μπορεί να είναι εδώ σήμερα, αλλά μου ζήτησε να τον εκπροσωπήσω για να μιλήσω για το θέμα αυτό. Αυτή είναι η δική μας γνωμοδότηση για την εφαρμογή της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα αρμόδια επιτροπή επί της ύλης είναι η Επιτροπή Περιβάλλοντος και προφανώς ε, εμείς ε, καλούμαστε να, να εισάγουμε μία νότα πραγματισμού και ρεαλισμού στο όλο θέμα. Είμαι τις αρμοδιότητες της Επιτροπής. Το σχέδιο των ε, προτάσεων, επτά συστάσεις έχει κάνει ο συνάδελφος, συμπεριλαμβάνοντας τα εγγραφά σας, καλύπτουν τη σημασία του να εστιαστούμε στους υδατρινούς πόρους, ε, στην καλύτερη διαχείρισή τους, στα πλαίσια του προγράμματος ορίζοντας 2020, αυτό αποτελεί την προτεραιότητα και καλεί την ε, πολιτική για την έρευνα να ανταποκριθεί στους προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Γεωργία σημειώνει ότι όλες οι επιχειρήσεις εξαρτώνται από τους υδάτινους πόρους και αυτό θεωρώ ότι είναι αλήθεια. Όλοι εξαρτώμαστε από το νερό. Πρόκειται για ένα απαραίτητο αγαθό στη ζωή και επίσης η βιομηχανία εξαρτάται από τους υδάτινους πόρους. Ζητά από την βιομηχανία και από την έρευνα να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις υφιστάμενες προκλήσεις με τον τρόπο αυτό. Απλά λέμε ότι θα πρέπει να σχεδιάσουμε πώ χρησιμοποιούμε το νερό, γιατί καθίσταται σπάνιο πόρος και μία από τις συνέπειες της κλιματική αλλαγής είναι η έλλειψη ύδατος σε κάποιες ε, χώρες, σε κάποια μέρη του πλανήτη και η... το πλεόνασμα υδάτων σε άλλα μέρη. Εδώ μου ζήτησε ο εισηγητής να σημειώσουμε ότι και η ανακύκλωση του ύδατος ε, θα παίξει σημαντικό ρόλο και ότι καλό θα είναι να καλύπτονται τα προγράμματα και ανάπτυξης. Ζητά καλύτερο συντονισμό επίσης και ανάπτυξη ευρωπαϊκών πολιτικών για τα ύδατα βάσει των σχεδίων διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών. Αυτό αποτελεί πραγματικά κάτι που εντάσσεται στα πλαίσια της κοινή λογικής και είναι σημαντικό για τη διαχείριση των υδάτων. Επισημάνει επίση τι δυνατότητε για καλύτερη διαχείριση των δεδομένων, βασιζόμενη στην ευελτίωση των συντηρητικών στοιχείων και στη χρήση, την περαιτέρω χρήση του προγράμματο GMES για να παρακολουθούμε καλύτερα την κατάσταση των υδάτων εμπόρων και των ε, αναγκών βελτίωσης αυτών. Σημειώνει τις δυνατότητες της υδραυλικής ενέργειας ως μορφή παραγωγής ενέργειας που είναι μηδενική σε άνθρακα και βασίζεται στους ίδιους πόρους αποκριθεί αποτελεσματικά στις απαιτήσει του Ευρωπαϊκού Ενεργειακού Ενεφοδιασμού και ζητά την ανάπτυξη νέων και ανατόμων ενεργειακών λύσεων στον αναλογό τομέα. Και αυτό γιατί μεγάλο τμήμα της υδραυλικής ε, των υδροηλεκτρικών πόρων έχουν ήδη αξιοποιηθεί. Θα πρέπει να είμαστε λοιπόν κοινωνικοί και αυτό αποτελεί προσωπικό μου σχόλιο ότι οι μικρές, τα μικρά εργοστάσια υδρολεκτικής ελέγχειας έχουν σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουν. Γιατί ξέρετε, το άθροισμα πολλών μικρών ε, εργοστασίων μπορούν να, έχουν, να έχει μεγάλο αποτέλεσμα παραπένει την Επιτροπή ο εισηγητής να αναπτύξει μια συνεκτική προσέγγιση της εσωτερικεύσης των δαπανών που απορρέουν από τη χρήση και τη μόλυνση των υδάτων Αυτό είναι σημαντικό. Ο κόσμος πρέπει να ξέρει ότι φυσικά το νερό είναι δωρεάν, αλλά η σύλλεξή του, η χρήση του, η ε, ο καθαρισμός του δεν είναι δωρεάν και τέλος. Ο κ. Ζημάνσκι ζητά την ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας με τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς με σκοπό τον αποτελεσματικό χειρισμό των υφιστάμενων προκλήσεων προκειμένου εκ νέου να βελτιωθεί η κατάσταση. Εφτά σημεία τα οποία σκοπεύει λοιπόν να υποβάλει τα οποία και συστήνω την Επιτροπή και ευχαρίστω να ακούσω τι έχουν να πούν και οι συνάδελφοι. Ευχαριστώ, συνάδελφε Ο συνάδελφο Φράγκο έχει το λόγο. Euh, Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Συγχαίρω τον εισηγητή για το σχέδιο γνωμοδότηση και τι ιδέε που προτείνει για την πρόκληση στο τομέα του ύδατο το θέμα του είδατο συζητείται στο τέλο του Παγκοσμίου Φόρουμ του Νερού που έγινε την περασμένη εβδομάδα στη Μασαλία. Είναι σημαντικό για το θεσμικό μα όργανο να συνεχίσει τον όλο προβληματισμό επί του θεματο Η διαχείριση των υδάτων είναι σημαντική πρόκληση που δεν έχουμε δικαίωμα να μελήσουμε. Διαπιστώνω ότι το νερό είναι ο φτωχό γείτονα τη περιβαλλοντική πολιτική, ενώ ο ρόλο του είναι ζωτική σημασία γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να θεσπίσει φιλόδοξη και ισχυρή νομοθεσία. Ήδη έχουμε κάνει σημαντικά βήματα, διότι το νερό αποτελεί μια από τι προτεραιότητε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Για το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο θα ήθελα να εμπλουτίσω το κείμενο σε διάφορου τομεί. Ε, στον τομέα τη γεωργία καταρχά, χρειάζεται να έχουμε μια ειδική προσέγγιση όσον αφορά το νερό. Οι ανάγκε σε ποιότητα και ποσότητα στον τομέα είναι διαφορετικέ και θα πρέπει να βελτιστοποιήσουμε τους πόρους ανάντι και κατάντι πρόκλησή μας είναι να έχουμε ένα λιγότερο λέμαργο σε πόρου σύστημα. Η λύση περνά μέσω της έρευνας, αυτό είναι σίγουρο. Στις τροπολογίες που προετοιμάζω θα ήθελα να επιμείνω επί της ανάγκης που υπάρχει για έρευνα και για καινοτομία για να αυξηθεί η ποιότητα, να ευνοηθεί η επεξεργασία και να βελτιστοποιηθεί η διανομή. Χρειαζόμαστε νέες τεχνολογίες και χάρη στην έρευνα θα βρούμε αυτές τις λύσεις μέσω της έρευνας ε, ενώ την τεχνολογία εχμής χωρίς να ρισμονούμε και τις πράσινες τεχνολογίες για να ευνοηθούν αυτές οι λύσεις θα πρέπει να υπάρχουν συστάδες ε, στην Ευρώπη μελέτης θεματικής. Στην παράγραφο 2 υπογραμμίζεται ρόλος κρίσιμος για την οικονομία από πλευράς ύδατος. Χρειάζεται διάφοροι φορείς βιομηχανικοί να εμπλακούν στην προσπάθεια και να εφαρμόσει συγκεκριμένα μέτρα για αποτελεσματική χρήση του νερού και επεξεργασία του. Ε, θα ήθελα να επιμείνω επί δύο θεμάτων. Πρώτα απ' όλα η ενεργειακή βιομηχανία. Η ενεργειακή βιομηχανία δραματίζει σημαντικό ρόλο στη διαχείριση του δικτύου των υδάτων, κυρίω μέσω υδρολεκτική ενέργεια. Τα χρησιμοποιημένα ύδατα είναι μια πηγή ενέργεια και αυτά που θα πρέπει να τα εκμεταλλευτούμε το ενεργειακό περιεχόμενο του ύδατος είναι κάτι πραγματικό, είναι δυνατό να αντλήσουμε ενέργεια μέσω ανάκτησης θερμότητας ή μέσω αξιοποίησης οργανικών υλών που μεταφέρει. Η βιομηχανία του τουρισμού. Ο τουρισμός παίζει ένα σημαντικό ρόλο στην ευρωπαϊκή οικονομία. Αυτό ισχύει στις ε, περιοχές κοντά στους ε, ποταμούς και στα ιαματικά ε, λουτρά και έχουμε και τις ακτές που γαλάζιας σημαίας θα πρέπει οι επαγγελματίε του τουρισμού να συμμετάσχουν στην προσπάθεια για να γνωρίσουν τι δυναμικό διαθέτουν και τι ευθύνε έχουν βέβαια να προωθηθούν οι βιώσιμε πρακτικές. Θα πρέπει, θα πρέπει να βαθύνουμε στο θέμα τη επεξεργασία των υδάτων. Χρειάζεται μια προσέγγιση διαφορετική από τη διανομή. Εκεί Εξαρτάται από πώ θα χρησιμοποιηθεί το νερό η βιομηχανία, την κατανάλωση. Θα πρέπει να διαφοροποιηθεί η προσέγγιση όσον αφορά την κατεργασία συναρτήση τη προελεύσεω του ύδατο προ ανάκτηση. Το θέμα τη προμήθεια εφοδιασμού θα πρέπει ε, να συνδεθεί με την ε, διαδικασία επεξεργασία. Επενδύσει. Πρέπει να επενδύσουμε στο νερό ακόμα και στην ήπειρό μα. Το χρειαζόμαστε για να αντιμετωπίσουμε τη λειψιδρία αλλά και για λόγους οικολογικούς Δύο εκατομμύρια Γάλλοι, μου λένε σήμερα, πίνουν νερό που δεν είναι κατάλληλο. Σημαντικές είναι επενδύσεις και σε κάποιες μητροπόλεις μέχρι 70% του διανεμούμενου ύδατος χάνεται λόγω διαρών του δικτύου τεράστιο το περιθώριο για βελτιώσεις και πρέπει να κάνουμε μεγάλες προσπάθειες να εφαρμόσουμε αποτελεσματική πολιτική για το νερό και θα πρέπει να μιλήσουμε γι' αυτό για διακυβέρνηση. Πρέπει να βρούμε την καλή λύση συνεργασίας μεταξύ ιδιωτικού τομέα, δημόσιου τομέα και χρηστών. Και εκεί θα υποβάλω σχετικέ τροπολογίες. Καταλήγοντας, συμφωνώ με τον εισηγητή για, την... πολιτική γειτονία και τη διεθνή συνεργασία. Πράγματι είναι σημαντικότατο. Οι στόχοι της χιλιετίας μας σωθούν προς σωστή κατεύθυνση καλώντας μας να προχωρήσουμε και πιο πέρα. Θα ήθελα να τονίσω όμως τη Μεσογειακή Λεκάνη ε, στα πλαίσια της ενώσεως της Ευρωμεσογειακής ε, Μεσογείου. Ενέκρινε ε, στη Γάζα πρόγραμμα αφαλάτωσης ύδατος η συνέλευση αυτή. Ασχολείται ο φορέας με το νερό, πρέπει να υποστηρίξουμε αυτή την αρχή. Θα πρέπει οι όμορες χώρες να συζητούν και να συνεργαστούν για το θέμα του νερού το νερό είναι φορέα ειρήνη ενδεχομένω να μην αμελούμε αυτή την ε, σημαντική πτυχή και σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Φράγκο. Ο κύριο Τζέρεκ έχει το λόγο. Ε, Τζέρεκ, ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε. Είναι πάρα πολύ θετικό. Πολύ θετικό ότι έχουμε ένα τέτοιο σημαντικό θέμα να ζητήσουμε, διότι χωρίς νερό δεν υπάρχει ζωή κυρίες και κύριοι το νερό είναι δημόσιο αγαθό και ακριβώς θα πρέπει να θεωρείται προσβάσιμο σε όλους, από όλους, ανεξαρτήτως εισοδήματος. Και άρα θα πρέπει να είναι ποιοτικό αυτό το δημόσιο αγαθό. Πρόκειται για μια επένδυση, μια δημόσια επένδυση και γι' αυτό και χρειάζεται μια βιώσιμη διαχείριση η υπόθεση των υδατίνων πόρων. Επίσης η ιδιωτικοποίηση της παροχή του ύδατο είναι ένα, αλλά δεν θα πρέπει να οδηγήσει στο, σε, σε καταστάσεις μονοπωλιακές. Να θεωρηθεί το νερό δημόσιο αγαθό. Κατά τρίτον, πάρα πολύ συχνά έχουμε συναγερμό για πλημμύρες. Ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι το οποίο απαιτεί κάποιες προσπάθειες ανάλυσης, διερεύνησης των αιτιών των πλημμυρών. Επίσης, θα πρέπει να μην παραλείψουμε να δούμε τι γίνεται και με τις γειτονικές μας χώρες. Και αυτό γιατί τα φράγματα δεν συμπίπτουν πάντοτε με τα σύνορα. Και τώρα εννοώ τα πολωνοουκρανικά σύνορα. Τώρα ε, η απερίμωση ε, έχει σημασία εν προκειμένου και έχουμε ακούσει ε, το τι γίνεται στην Ισπανία, στη δε χώρα μου, την Πολωνία επίσης. Έχουμε κάποια προβλήματα κι εμείς, άρα χρειάζεται να ληφθεί δράση και να γίνει κάποιο είδου ίδρυυση, πότισμα. Και θα πρέπει επομένως η Ευρωπαϊκή Ένωση επιγόντως να ασχοληθεί με αυτό το ζήτημα. Οπότε θα πρέπει να αναζητηθούν πόροι από το Ταμείο Συνοχής. Και αυτοί οι πόροι να χρηματοδοτήσουν τις ε, υποδομές με τρόπο καλύτερο από ό,τι μέχρι σήμερα. Όλοι οι πόροι μέχρι σήμερα πάντως πηγαίνουν στη, στην κατασκευή δρόμων και πόρα πολύ λίγα για τα ύδατα. Οντί. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρώτα πρώτα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για το έργο που επετέλεσε και επίση ε, συμφωνώ με τα όσα είπε ο προλαλής σας συνάδελφος. Ε, να σας πω τις δικές μου σκέψεις τώρα. Νομίζω ότι με δεδομένη την δημογραφική τάση στον πλανήτη μας θα πρέπει να ασκήσουμε μια ευρωπαϊκή πολιτική για τα ύδατα. Έχουμε πολύ ήλιο, αλλά έχουμε και ε, πάρα πολύ ίδρυυση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γύρω-γύρω έχουμε πολλές θάλασσες και ωκεανούς. Και επομένως είναι αδιανόητο να μην μπορούμε να αξιοποιήσουμε αυτόν όλο τον πλούτο και να είναι κινητήρια δύναμη ε, αυτή, αυτό το πλεονέκτημά μας. Έχουμε 800.000 ανθρώπους που δεν μπορούν να έχουν νερό. Ε, πρέπει να γίνουν γεωτρήσεις, θα πρέπει να δώσουμε το παράδειγμα, γιατί πολλές φορές γίνεται πόλεμος πραγματικός για το νερό και σκοτώνει ένα τον άλλο. Τώρα, όσον αφορά τη δική μας Ήπειρο, ήρθε η ώρα να μελετήσουμε αυτήν την οδηγία για το νερό. και στη δική μου περιφέρεια υπάρχει ε, το ζήτημα των, των, λιμνών οι οποίες είναι υποτιμημένες γιατί υπάρχουν περιορισμοί όσον αφορά τη διαχείριση του ύδατος από πλευράς οικολογικής, περιβαλλοντικής ε, πολιτικής. Και επίσης υπάρχει και ένα ζήτημα με, με, τα, με, με τα ψάρια που ζουν στο γλυκό νερό και να σταματήσει να υπάρχει η αποθάρρυνση, τα αντικίνητρα αυτής της ε, οδηγίας για τα ύδατα. Ε, άλλο στοιχείο τώρα, σε σχέση με τις υποδομές, διαπιστώνεται ότι υπάρχει πρόβλημα νερού στην Βαργελόνη. Υπάρχει επίσης θέμα ε, ε, αυτών των, τελών που καταβάλλονται για τον ε, Ρήνο, αυτό το τεράστιο ποτέ που είπε και ο συνάδελφος ε, Φράγκο. Και τα σχετικά προγράμματα επίσης έχουν μπλοκαριστεί από περιορισμούς περιβαλλοντικούς για να προστατευτεί ξέρω ο μπλε καραβέο και πράσινη ράχνη. Άρα χρειάζεται κάποιο είδου σχεδιασμό πολιτικό για την υποδομή για τα υδατά. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μελετήσει μία, έναν, φορέα. Ένα φορέα που να έχει την κυριότητα όλων των σχετικών υποδομών και επομένως να εξυπηρετούνται όλοι οι Ευρωπαίοι παντού, σε όλη την Ευρώπη, με με πρόσβαση στα νερά ε, από όπου και αν προέρχεται το, νερό και να υπάρχει επίσης και η δέουσα έρευνα, το πρόγραμμα έρευνας. Γιατί θα έπρεπε να είμαστε πρωτοπόροι όσον αφορά τις πολιτικές ε, του είδατος. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να τοποθετηθεί, να δείξει η πολιτική βούλη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να είμαστε παράδειγμα προς μίμηση όσον αφορά τα είδατα ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ Ο κύριος Κέλλη Ευχαριστώ πολύ. Πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Το νερό όπω και ο αέρα είναι δύο πόροι άνευ των οποίων δεν μπορούμε να ζήσουμε και θεωρούμε ως δεδομένα. Και θέλω να συγκεντρωθούμε στο θέμα. Και στη χώρα μου που βρέχει πολύ ο κόσμο θεωρεί ότι πρέπει να είναι τζάμπα το νερό να δίνεται και να προτείνουμε να μετρηθεί το νερό και να πληρώσει το νερό είναι κάτι το οποίο του ενθουσιάζει, αλλά νομίζω ότι είναι αναγκαίο. Διότι θα το εκτιμήσουν καλύτερα, πιστεύω. Και θα το χρησιμοποιούν καλύτερα. Δεν το χρησιμοποιούν τόσο για να πλύνουν τα αυτοκίνητα και να ποτίζουν και να το σπαταλάνε. Αυτό που είπε και ο Στίτσεστερ τώρα, όσον αφορά την υδροελεκτρική ενέργεια, είναι πολύ σημαντικό. Είναι ένα τομέα που δεν έχουμε συζητήσει επαρκώς όταν μιλάμε για τις ανανεώσιμες πηγές ενεργείας. Ας το συζητήσουμε τώρα και η μικροπαραγωγή ενέργειας από ηλεκτρική ενέργεια είναι κάτι που θα μπορούσε να εξεταστεί. Η ανακύκλωση του νερού είναι κάτι που πρέπει να ενθαρρυνθεί. Ετέθηκε το θέμα του τουρισμού σε σχέση με το νερό. Έχετε σκεφτεί πόσα πανδοχεία, ξενοδοχεία, αν πόσα ξενοδοχεία και πανδοχεία αναμειγνύονται σε αυτό. Και πόσο νερό χρησιμοποιείται χωρίς να χρειάζεται. Χρειάζεται παιδεία, εκπαίδευση όσον αφορά τη σπατάλη του νερού. Και πρέπει να γίνουν πιο υπεύθυνοι οι πολίτες. Χρειάζεται αύξηση της ευαισθητοποίησης. Χρειάζεται παγκόσμια προσέγγιση αλλού σπανίζει το νερό, αλλού υπάρχει περισσότερο νερό. Πρέπει να έχουμε σφαιρική εικόνα. Να σκεφτούμε και κάτι άλλο. Διαρροές νερού από τους σωλήνες. 70% είπε κάποιος. Στη χώρα μου υπολογίστηκε 50% του νερού τη χάνεται. Αυτό είναι σπατάλι. Και αυτό θα πρέπει να αντιμετωπιστεί το ταχύτερο δυνατό. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ Κυρία Κέλλη, ο συνάδελφος Ρούμπικ έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι το δίκαιο για τα υδάτα μας δίνει μεγάλες ε, ευκαιρίες σε ό,τι αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και νομίζω ότι για τις υπηρεσίες περιβάλλοντος και για όλες τις άλλες υπηρεσίες στα θέματα διαχείρισης του ύδατος είναι ε, πολύ σημαντικό να σκεφτούν στρατηγικέ αμοιβαίω υποφελεί. Πώ μπορούν να συνδυαστούν δηλαδή τα οικολογικά ζητήματα με τα οικονομικά ζητήματα. Για παράδειγμα, στην ε, οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα, σε ό,τι αφορά τα αποθέματα εχθείων, Ποιε δυνατότητε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για συνδυασμό τεχνολογικών πρακτικών, για την βέλτιστη πρακτική των υδάτων για ανανεώσιμε ενέργειε, αλλά παράλληλα βέλτιστη ε, διαμόρφωση των περιβαλλοντικών όρων. Νομίζω λοιπόν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει μείνει λίγο πίσω στο σημείο αυτό σε ό,τι αφορά τεχνολογικές μελέτες αντικτύπου, οι οποίες θα καταδείξουν τι εναλλακτικέ υπάρχουν για τους παραγωγούς ε, εναλλακτικών ενεργειών και αφενός να βελτιωθεί η οικολογική κατάσταση, αλλά αφετέρου να μην σπαταλάτε άσκοπα νερό. Νομίζω ότι στο σημείο αυτό θα ήταν απαραίτητη μια πρωτοβουλία για το πώς θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε το 100% των υδάτων για υδρολεκτικά εργοστάσια, αλλά και σε ποταμούς, να μην χρησιμοποιούνται μόνο οι παραδοσιακές τεχνικές λύσεις, αλλά και νέες καινοτόμες λύσεις. Πώς μπορούμε όλα αυτά να τα εγγυηθούμε. Τελευταίο σημείο, χρειαζόμαστε κατεπηγόντως και τα εργοστάσια όσμωσης. Μια χημική διαδικασία για τα α, ύδατα. Θα μπορούσαμε στο σημείο αυτό να δούμε πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το μείγμα αυτό θαλάσσιων και μη υδάτων για να τις πηγές ενέργειας σε ό,τι αφορά υπόγεια ή τα οποία καταλήγουν για παράδειγμα στη θάλασσα και αυτό νομίζω αποτελεί ένα σημαντικό θέμα που παρουσιάζει ευκαιρία για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να φροντίσει η τα οποια καταληγουν για παραδειγμα στη θαλασσα και αυτο νομιζω αποτελει ενα σημαντικο θεμα που παρουσιαζει ευκαιρια για να τις πηγες ενεργειας εδω λοιπον θα πρεπει να φροντισει η επιτροπη να καταρτιστεί ένας κατάλογος με συγκεκριμένα σημεία προκειμένου να δούμε ποιες είναι οι προτεραιότητες που θα πρέπει να τεθούν για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και επίσης να σημειωθεί τι θα πρέπει να γίνει σε περίπτωση που είναι απολύτως απαραίτητο. Ευχαριστώ. Τελείωσαν οι παρεμβάσεις. Δίνω το λόγο στον Πασκάν Αντιγιού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Α, δεν είναι εδώ. Ο εισηγητή έχει το λόγο λοιπόν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και τους συναδέλφους για τις ε, συνεισφορές τους. Προφανώς ε, σημείωσα τα σχόλιά σας. Ελπίζω να μπορέσει να τα διαβάσει ο συνάδελφος Σιμάνσκι και προφανώς οι συνάδελφοι έχουν σκεφτεί το θέμα αυτό και το πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τη διαχείριση των υδάτων. Όλοι συμφωνούμε ότι πρόκειται για ένα πολύ πολύτιμο αγαθό για τη ζωή μας και για τον τρόπο ζωής μας. Να ευχαριστήσω τον κύριο Φράνκε για τη, τις πολλαπλές του προτάσεις που είναι νομίζω ενδεικτικές της σημασίας του θέματος. Δεν θα τις διατρέξω όλες. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό ο κατάλογος των ιδεών που ακούσαμε. Θα ήθελα ωστόσο να αναφέρω το θέμα των απολειών κατά τις μεταφορές. Και άλλοι συνάδελφοι το ανέφεραν. Προφανώς, σε ένα πιο εξελιγμένο δίκτυο το οποίο όπως αυτό που έχουμε στην Ευρώπη και στα κράτη-μέλη, δεν είναι αποδεκτό να υπάρχουν τόσο, μεγάλα, τόσο μεγάλο όγκος απολειών. Από την εμπειρία μου στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου η αγωγή είναι 100-150 χρόνων σε πολλές περιπτώσεις. Δεν ε, είναι περίεργο το ότι δείχνουν την ηλικία τους και άρα λοιπόν υπάρχει μεγάλη ανάγκη για επενδύσεις στις υποδομές και επειδή η αγωγή αυτή είναι υπόγειη δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι ο κόσμος δεν τα αντιλαμβάνονται αυτά τα πράγματα απαραίτητα σε ό,τι αφορά δηλαδή όλες αυτές τις διαρροές. Αλλά κοιτάξτε, πρόκειται για ένα αρκετά απλό και βασικό τρόπο διαφύλαξης του πόρου. Κύριε Γκέρεκ, δεν σας ικανοποιεί αν κατάλαβα καλά οι διατάξει ε, για τον κλάδο σε ό,τι αφορά τις διατάξεις για τον δημόσιο κλάδο. Αυτό σε πολλές περιπτώσεις ισχύει. στον Ηνωμένο Βασίλειο και πάλι να αναφερθώ, διαπιστώσαμε ότι διακρίνονται, ε, κάνοντας μάλλον ένα διαχωρισμό την παροχή νερού, από την, της παροχής νερού από τις άλλες ε, δημοτικές υπηρεσίες και ιδιωτικοποιώντας με ωστόσο ε, αυστηρή νομοθεσία την ιδιοκτησία αυτή, διαμορφώνονται μεγάλη αποτελεσματικότητα στη διαχείριση. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για την αντιμετώπιση τέτοιων απολειών ακριβώς σε ό,τι αφορά τα ανατοτά όρια τιμών, σε ό,τι αφορά τις προδιαγραφές που χρειάζονται για επένδυση στις υποδομές. Άρα ένα σύστημα σύμπραξης ιδιωτικού και δημοσίου τομέα νομίζω ότι θα, έχει τη δυνατότητα να λειτουργήσει Καλά, δεν θα ήθελα να το αποκλείσω και συμφωνώ με τον κύριο Οντή για το θέμα πρόσβασης στο νερό σε περίπτωση που ο κόσμος δεν έχει νερό. Αυτό θα σήμαινε αποτυχία της βιομηχανικής κοινωνίας και θα έπρεπε κατεπηγόντως να αντιμετωπιστεί γιατί δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι όλοι χρειάζονται το νερό. Καταλαβαίνω το επιχείρημα για μια πανευρωπαϊκή προσέγγιση. Το πρόβλημα ωστόσο είναι το εξή ότι έχουμε τα συστήματα βάση ποταμών και δεν νομίζω ότι κανείς έχει εθνικό δίκτυο παροχής ύδατος. Θα πρέπει να αποτεχτούμε ότι το κόστος που θα σήμαινε η δημιουργία ενός εθνικού ή πανευρωπαϊκού δικτύου υδροδότησης θα ήταν τεράστιο, τεράστιο το κόστος επενδύσεων σε ό,τι αφορά θέματα για διασύνδεσης, ε, αναβάθμιση των αγωγών. Άρα θεωρώ ότι είναι θεμητός ο στόχος κατάργησης των ανισοτήτων. Όλοι τα γνωρίζουμε. Στη χώρα μου σε άλλα μέρη έχουμε ξηρασία, σε άλλα μέρη έχουμε πλημμύρες, το οποίο είναι δύσκολο να το κατανοήσει κανείς ίσως, αλλά είναι γεγονός. Να ευχαριστήσω τους συναδέλφους λοιπόν και θεωρώ ότι οι προτάσεις του κυρίου Ρούμπιχ για το να επανεξεταστούν οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στην διαχείριση των υδάτων είναι πάρα πολύ θετικό. Και αυτό νομίζω εντάσσεται σε αυτό που ανέφερε ο κύριος Σιμάνσκι για τη σημασία της έρευνας. Μπορεί να θεωρούμε ότι το νερό και η ίδρυυση είναι κάτι απλό, και ξεκάθαρο, αλλά πολλά μπορούν να γίνουν σε ό,τι αφορά την έρευνα, την καινοτομία, για την εκμετάλλευση και την διατήρηση της καθαρότητας, αν θέλετε, των υδάτων. Έχω λοιπόν σημειώσει πολλές σκέψεις, θα τις διαβιβάσω στον κύριο Σιμάνς και σας ευχαριστώ και προσβλέπεις τις τροπολογίες που θα καταθέσουν οι συνάδελφοι. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ συνάδελφε Τσίτσεστερ. Να σας πω ότι η προθεσμία για τις τροπολογίες είναι 5η 12 Απριλίου, 12 το μεσημέρι. Πάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Η Κριστίνα Ζούμπερ θα μας μιλήσει για τα ευρωπαϊκά προγράμματα για τις ε, κοινωνικές αλλαγές, για την κοινωνική αλλαγή και την καινοτομία. Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αυτός ο κανονισμός που προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει σαν στόχο την δημιουργία ενός προγράμματος. Είναι ένα πρόγραμμα που θα έχει σαν στόχο την κοινωνική αλλαγή και την καινοτομία κυρίως όσον αφορά την απασχόληση και τα συναφή θέματα. Βασίζεται επί τριών προγραμμάτων του Progress, του Eurest και του Ευρωπαϊκού Εργαλείου για τη Μικροχρηματοδότηση που δημιουργήθηκε το 2010. Πάνω σε αυτούς τους τρεις άξονες εδράζεται. Εξετάζοντας το μέσω ήτρε που το εξετάζουμε βάσει της γνωμοδοτήσεως πρέπει να πούμε ότι σχετίζεται πολύ με τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Θέλω να εστιαστώ επί τριών σημείων της γνωμοδοτήσεως. Πρώτα απ' όλα, πρόσβαση στις πιστώσεις για τις μικροεπιχειρήσεις. Πιστεύουμε ότι η πίστοση που προσφέρεται στις μικροεπιχειρήσεις, κυρίως κατά μία περίοδο προβληματική με μεγάλη ανεργία που επικρατεί στην Ευρώπη σημαίνει ότι δεν πρέπει μόνο να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε αυτές τις μικρό επιχειρήσεις αλλά θα πρέπει να προσπαθήσουμε να τις ενθαρρύνουμε και να τις βοηθήσουμε να προσαρμοστούν στις νέες αναδυόμενες τεχνολογίες αυτό είναι σημαντικό αν θέλουμε να εγγυηθούμε την ύπαρξη ρευστότητας και την ανεξαρτησία. Να τις προστατεύσουμε από τις μεγάλες επιθετικές ε, εταιρείες. Το θέμα της τεχνολογικής καινοτομία είναι σημαντικό για την ανταγωνιστικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των μικρό επιχειρήσεων. Άλλο θέμα είναι το εξής η δημιουργία θέσεων απασχόλησης θα πρέπει να σχετιστεί με την αλλαγή δεξιοτήτων, να σχετίζεται με πολιτικά θέματα, κοινωνικά θέματα, βιομηχανική πολιτική. Πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας το θέμα της εφιούς χρήσεως των πόρων και ε, των χαμηλών εκπομπών ε, ενώσεων του άνθρακα. δοθέντων των προβλημάτων των δημιουργωμένων από την ανεργία στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή θα πρέπει να φροντίσουμε το ώστε το θέμα της χρηματοδότησης της μικροχρηματοδότησης και των κοινωνικών επιχειρήσεων να μην μειωθεί, να το αυξήσουμε, να το πάμε στο 30%. Έτσι θα, δημιου... θα βοηθείται η δημιουργία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Να συστήνονται και δημιουργούνται μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ευχαριστώ. Ο συνάδελφος Ρούμπιχ έχει το λόγο. Ευχαριστώ, συνάδελφε. Νομίζω ότι η κοινωνική διάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η κοινωνία ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την ανεργία στο μέλλον, θα διαδραματίσει ιδιαίτερο ρόλο. Κοιτώντα ότι ιδιαίτερα οι νέοι είναι αυτοί που πλήττονται ιδιαίτερω από την ανεργία, διαπιστώνουμε ότι πρέπει να καταβάλουμε πιο πολλές προσπάθειες προκειμένου οι νεαροί επιχειρηματίες να λάβουν κίνητρα. προκειμένου οι εργοδότες μαζί με τους εργαζομένους να πετύχουν υψηλούς μισθούς για υψηλή εξειδίκευση. Και ιδιαίτερως να προωθήσουμε τις νεαρές επιχειρηματίες. Θα πρέπει λοιπόν να κοιτάξουμε στην έκθεση μήπως τα κοινωνικά δικαιώματα τα οποία ε, θα πρέπει να έχουν οι νεαρές επιχειρηματίες να είναι τα ίδια με αυτά που αναλογούν και στους αντίστοιχους επιχειρηματίες αρσενικού φύλου. 85% των θέσεων εργασία ξέρουμε, προκαλούνται, μάλλον προέρχονται από νέες επιχειρήσεις. Αλλά για την ε, νέα γυναίκα, ο κίνδυνος που ε, περιέχεται για την ίδρυση νέες επιχειρήσεις είναι και προσωπικός, αλλά και σε ό,τι αφορά το ιδιωτικό κεφάλαιο. Όλα αυτά θα πρέπει να αποτυπώνονται και στους μισθούς. Θα πρέπει λοιπόν να είναι ανάλογοι οι μισθοί και να υπάρχει και ένα πριν κινδύνου. Και να υπάρχει ασφαλώς και μία, ένα επιτόκιο στο κεφάλαιο το οποίο έχει ε, επενδυθεί. Αυτά τα τρία στοιχεία λοιπόν αποτελούν τη βάση για το επιχειρήν. Και φυσικά τι γίνεται με τους νεαρούς επιχειρηματίες οι οποίοι αποτυγχάνουν, που δεν παίρνουν για παράδειγμα, δεν κερδίζουν τον διαγωνισμό. Ποια είναι η κοινωνική τους εξασφάλιση, ποια κοινωνική εξασφάλιση θέλουμε να έχουν στο μέλλον. Και νομίζω ότι χρειάζεται τουλάχιστον ε, στο εργατικό δίκαιο μία υποσημείωση για την κοινωνική ασφάλεια αυτών που τολμούν να γίνουν νέοι επιχειρηματίες. Και εδώ πέρα θα πρέπει να μας παρουσιάσει μία έκθεση πρωτοβουλίας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το τι γίνεται στην περίπτωση που αποτυγχάνει ο νεαρός επιχειρηματίας. Πώς τοποθετείται και πώς αντιμετωπίζει η κοινωνία τους νεαρούς επιχειρηματίες στο, στην περίπτωση αυτή. Γι' αυτό λοιπόν χαίρομαι ιδιαίτερα που έχετε θέσει το θέμα αυτό σήμερα στην ημερήσια διαταξή. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ, συνέφερε Ρούμπικ. Δεν υπάρχει άλλος που θέλει να μιλήσει. Το λόγο τον έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Euh, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σε όλους τους βουλευτές. Εγώ τώρα θα τοποθετηθώ σε κάποια από όσα ανέφερε ο εισηγητής, δηλαδή η πρόσβαση στην ε, τραπεζική πίστοση για τις μικροεπιχειρήσεις, δημιουργία θέσεων απασχόληση και σε ποιο βαθμό μπορεί να βοηθήσει αυτό το νομοθέτημα. Επίσης, ε, εν τέλει θα σας ε, μιλήσω για την ανεργία και για το πώς είναι δυνατόν να βοηθήσουμε με το νομοθέτημα στην καταπολέμηση του φαινομένου αυτού. Τώρα, όσον αφορά το πρώτο σημείο, όσον αφορά, έλεγα, την πρόσβαση στις πιστώσει για τις μικροεπιχειρήσει πρόκειται για μία από τι δραστηριότητε, τι οποίε προτείνονται από αυτό το νομοθέτημα και συγκεκριμένα εκεί που λέει ε, ε, κοινωνική πληγματικότητα κλπ. λοιπά Και επομένως ε, είναι ένας αυτό από του στόχους του νομοθετήματο. Οπότε θα πρέπει να είναι συμπερίληψη κοινωνική και προσβασιμότητα για τους μη προνομιούχους. Ε, έχουμε και στόχο ευρωτεριότητα άλλη ε, ε, όσον αφορά την ε, ίδρυση των ΜΜΕ και όσον αφορά την ίδρυση αυτών έχουμε άλλα νομοθετήματα στα πλαίσια του κοινοτικού δικαίου εν προκειμένου δεν υπάρχει ο στόχος να εξυπηρετηθεί αυτή η υπόθεση των νέων επιχειρήσεων. Επίσης έχουμε σχετικές τροπολογίες. Αυτές οι τροπολογίες αλλάζουν την, την εστίαση αυτού του νομοθετήματος όσον αφορά τις ΜΜΕ. Εμείς θεωρούμε ότι έτσι θα υπάρξει επικάλυψη με τα άλλα νομοθετήματα. Ε, συγκεκριμένα υπάρχει ένα νομοθέτημα για τις ε, ιδρύσεις των ΜΜΕ ως τα πλαίσια των δημοσιονομικών προοπτικών. Όσον αφορά τώρα τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, εδώ πέρα υπάρχουν δυνατότητες και με αυτό το πρόγραμμα θα μπορέσουμε να δούμε, να επισημάνουμε με μελέτες, με κάποια, ε, κάποιες κινήσεις που προτείνονται εδώ, το πώς θα βοηθηθεί η ανάπτυξη πράσινης της εργασίας ή λευκές της εργασίας όσον αφορά τον τομέα της πληροφορικής στα πλαίσια αυτού του προγράμματος και πιο συγκεκριμένα εκεί στην πτυχή λέει πρόοδος, ε, μπορούμε να βρούμε τέτοιες δραστηριότητες. Και έχουμε τώρα αυτά τα οποία είπε ο εισηγητής όσον αφορά ε, τους ε, τομείς με μεγάλων δυνατοτήτων και για το πώς μπορούν αυτές να αναπτυχθούν. Επίσης, πρέπει να σας πω ότι έχουμε εδώ πέρα άμεση διαχείριση με κάποια ποσά σχετικά μικρά σε σχέση με άλλα νομοθετήματα όπως το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Εν προκειμένου έχουμε το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης που προβλέπουν πολύ μεγάλες προοικοδοτήσεις όσον αφορά την προώθηση ανάπτυξη τέτοιων δραστηριοτήτων. Οπότε εδώ γίνεται μια σημαντική διάκριση μεταξύ αυτού του, μικρού εργαλείου σε επίπεδο κοινοτικό για αυτές τις προτάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο και από την άλλη μεριά έχουμε κάποια άλλα μέσα σε εθνικό επίπεδο. με μεγάλες προκατακτήσεις. Άρα δεν θα πρέπει να συγχαίουμε, να ανακατεύουμε αυτά τα μέσα. Είναι αυτό με μικρή εμβέλεια. Γιατί υπάρχουν και άλλα μεγάλες εμβέλειες όπως το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης που μπορούν να κάνουν πολύ περισσότερα για να προαγάγουν αυτόν τον τομέα δραστηριότητας. Τέλος, για να ολοκληρώσουμε όσον αφορά την ανεργία αλλά και τους διαθέσιμους πόρους και την πρόταση να αναθεωρηθεί το ποσοστό των διαφορετικών αξώνων του προγράμματος πρόκειται για ένα πρόγραμμα το οποίο όπως είπε η εισηγήτρια, η εισηγήτρια τρεις διαφορετικούς άξονες οι οποίοι όμως συνδυάζονται πρώτα-πρώτα το υπάρχον μέσο, progress και τώρα το ΕΡΕΣ για, την, για τη διευκόλυνση, ε, για την κοινωνική επιχειρηματικότητα προτείνει μια τροπολογία εισηγήτρια ώστε να τροποποιηθεί η πτυχή που αφορά δύο από αυτούς τους άξονες και λέει να συρρυκνωθεί το προγκρές και να αυξηθεί ε, ο άξονας μικροχρηματοδότησης σε σχέση με τη δική μας πρόταση. Θέλουμε να εξασφαλιστεί μία συνέχεια και προτείνουμε κάποιες προσαρμογές, κάποιες καινοτομίες όσον αφορά την ε, κατανομή των διαφορετικών κομματιών του μέσου σε σχέση με την σημερινή κατάσταση. Έχουμε επίσης την πρόταση της συγγήτριας να συρρυκνωθεί ο ένας άξονας και να ωφεληθεί να μεγαλώσει ο άλλος, αυτό βεβαίως και θα οδηγούσε ε, στην, στον αποκλεισμό κάποιων δραστηριοτήτων από το πρόγραμμα Progress. Και από δική μας πλευράς αυτό δεν είναι η πιο δόκιμη προσέγγιση, γιατί διαπιστώθηκε ε, όσον αφορά τη μέσοπρόθεσμη ε, αξιολόγηση του Progress. Πρόκειται για κάτι πάρα πολύ χρήσιμο και αποτελεσματικό. Αυτή η μεσοπρόθεσμη αξιολόγηση σας κοινοποιήθηκε συγκεκριμένα στην Επιτροπή σας της Απασχόλησης και μπορεί όποιος θέλει και η συγκήτρια να την συμβουλευτεί. Γιατί έτσι με πάρα πολύ λεπτομερή τρόπο αναδεικνύει ποια είναι τα υπέρ ε, τα πλεονεκτήματα του προγκρές και επομένω δικαιολογεί αυτό που θέλουμε δηλαδή να διατηρηθεί η πρικοδότηση. Α, και κάτι άλλο ότι η κυρία Συγγεντρία είπε ότι υπάρχει περιπλοκότητα σε αυτό το εργαλείο, αυτό το μέσο, γιατί συνδυάζει ε, τρία διαφορετικά μέσα που υπάρχουν. Εμεί, όμως θεωρούμε ότι αποτελεί απλούστευση. Αυτά τα, αυτά τα τρία νομοθετήματα, αυτά τα τρία ε, μέσα πολιτικής είναι παρόμοια. Είναι του τύπου άμεση διαχείριση, επίπεδο νοσιακό. Και αν επομένω τώρα τα ενοποιήσουμε θα είμαστε πιο αποτελεσματικοί και για όσο από εσά είσαστε κάπως εξοικειωμένοι θα προσέξατε ότι πέραν του κοινού στόχου πολλές φορές ε, έχουμε πάρα πολύ παρόμοιες διατάξεις. Άρα πρόκειται εδώ περί απλουστεύσεως και όχι περί ε, περισσότερης ε, περιπλοκότητας. Σας ευχαριστώ. Και κάτι θέλει να πει ο συνάδελφος Οντύπη να ολοκληρώσουμε. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Δεν συνηθίζεται αυτό, συγγνώμη. Πρόκειται περί αντιδράσεω μετά τι παρεμβάσει κυρίω Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή α, να κάνει την απλούστευση είναι καλά μαντάτα, είναι τα καλά μαντάτα τη ημέρα. Εγώ έχω κάποια αντίδραση. Θεωρώ ότι ο τίτλος του κανονισμού, πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως για την κοινωνική αλλαγή και την κοινωνική καινοτομία, σε σχέση με το περιεχόμενο, σαν πωλήσει, σαν, σαν του λαού, θεωρώ ότι υπάρχει διαφορά. Μιλάμε για 2 δισεκατομμύρια ε, ευρώ, μιλάμε για το Progress, το ΕΡΕΣ, για τρία εργαλεία, δεν τα ξέρει κανένα. Α αποφύγουμε ε, τον πολλαπλασιασμό όλων των συνθημάτων, διότι κάποια στιγμή ε, θα χαθούμε και θα πετύχουμε τα αντίθετα. Εγώ ήθελα να μιλήσω για έναν ορισμό που με ανησυχεί. Άρθρο 2. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει τον ορισμό μιας κοινωνικής επιχείρησης. Ας το συζητήσουμε αυτό. Κοινωνική επιχείρηση είναι μια επιχείρηση και ανεβάζω που έχει σαν στόχο κοινωνική επίδραση παρά τη δημιουργία κέρδους για τους ιδιοκτήτες ή τους εταίρους. Αυτό αναφέρει το κείμενο. Εδώ εισάγουμε ένα θέμα προς συζήτηση. Όλοι έχουμε συμφωνήσει, όσοι πολιτικές ομάδες επί της ιδέας επεξεργασίας της κοινωνικής οικονομίας αγοράς και μας εξηγεί τη διαφορά μεταξύ εμείς επιχειρήσεων που θα είναι κοινωνική όπως αποκαλείται και άλλων επιχειρήσεων που θεωρούνται κερδοφόρες. Εγώ δεν δέχομαι αυτού του είδους τους ορισμούς. Προσθέτω ότι τέσσερι γραμμές μετά λέμε ότι αυτέ οι κοινωνικές επιχειρήσεις υπόκεινται σε διαχείριση υπεύθυνη και διαφανή, που αυτό που θα σημαίνει ότι άλλες επιχειρήσεις οι κερδοφόρε των εισαγωγικών, δεν είναι ε, ούτε υπεύθυνε ούτε διαφανής. Πρέπει να προσέχουμε αυτό το διαχωρισμό μεταξύ επιχειρήσεων κοινωνικών όπως ορίζονται εδώ. Είναι αδέξιο να εισάγουμε αυτή την έννοια και έχουμε έννοια στα κράτη-μέλη όπως το δικό μου να μιλάμε για κοινωνική οικονομία, όχι για κοινωνική επιχείρηση. Και στην κοινωνική οικονομία που αναφέρουμε, όλες, όλοι οι οικονομολόγοι συμφωνούμε ότι βάζουμε τις διάφορες ενώσεις, τα ιδρύματα συνεταιρισμούς. Η Credit Agricole, παραδείγματο χάρη, είναι μεγάλη γαλλική τράπεζα. Είναι συνεταιρισμό που εξυπηρετεί του πελάτε. Αυτό που λέτε ότι εκεί συμμετέχουν οι πελάτε, ε, οι μέτοχοι κλπ. Ε, Συνεταιρισμού καμιά φορά είναι μισθωτοί και οι πελάτε. Αυτό τα καταλαβαίνουμε. Αυτό που λέμε είναι η οικονομία κοινωνική. Αλλά η κοινωνική επιχείρηση όπω την ορίζετε εδώ πέρα δεν νομίζω ότι θα οδηγήσει σε λύση. Θα το συζητήσουμε μεταξύ μα θα δημιουργήσει διαφορίες, χρειάζεται, διαφορές, χρειάζεται περαιτέρω συζήτηση αυτός ο όρος κοινωνικής επιχείρησης. Ευχαριστώ. Τσούμπερ, ο επόμενος θέλει να μιλήσει. Η επόμενη μάλλον. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να διευκρινίσω κάτι. Συμφωνούμε ότι το Progress είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Όπως κατέδειξε αυτή η αξιολόγηση. Όμως, εν ώψη του ότι λόγω της κρίσης αυξάνεται η ανεργία, θα πρέπει να γίνει μια νέα κατανομή των πόρων. Έχουμε λάβει υπόψη τη γνώμη των συναδέλφων και όλα αυτά θα τα ξανασυζητήσουμε για την ίδια γνωμοδότηση. Σας ευχαριστώ. Να σας ενημερώσω ότι η προθεσμία της τροπολογίας 5η 12 Απριλίου 12 το μεσημέρι. Συνάδελφος Κόβατς έχει τώρα το λόγο όσον αφορά τη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Ρωσία σχετικά με το εμπόριο εξαρτημάτων κατασκευαστικών στοιχείων μηχανοκινήτων οχημάτων. Σα ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Πρώτα πρώτα θα ήθελα να αρχίσω με το ότι οι επενδυτές θέλουν να κατασκευαστεί αυτοκινητοβιομηχανία στην Ρωσία και έχουν συρρυκνωθεί οι φόροι και δεσμοί από τα εξαρτήματα και έτσι προσπαθούν να συμμορφωθούν με τα όσα προβλέπονται για να συγκρατήσουμε τώρα την μετεγκατάσταση των επιχειρήσεων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε κάποιο είδους διαπραγματεύσεις με τη Ρωσική Ομοσπονδία. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό λαμβάνει υπόψη. Αυτό, αυτό είναι το θέμα της πρότασής μας για ανταλλακτικά, για εξαρτήματα, για ε, αυτοκίνητα για να μην έχουμε σύγνωση των ε, εισαγών γιατί αυτό το οποίο θέλουμε είναι αν έχουμε μείωση της, ε, των εισαγωγών τότε η Ρωσική Ομοσπονδία θα πρέπει να επιτρέψει την εισαγωγή των ανταλλακτικών αυτών και εξαρτημάτων ανάλογα με το πόσο θα μειωθούν οι εισαγωγές των ευρωπαϊκών εξαρτημάτων και ανταλλακτικών. Έχουμε 3% μείωση των εισαγωγών από την Ένωση. Τα συμβαλώμενα μέρη πρόκειται να υποπτεύσουν τα στατιστικά τα οποία υποβάλλονται κάθε Μάρτιο, το Μάρτιο για τις εξαγωγές και σύμφωνα με το άρθρο 10 η Ρωσική Ομοσπονδία πρόκειται να παράσχει στατιστικά εμπορικά δεδομένα. Με αυτή την συμφωνία θα εφαρμοστεί ό,τι συμφωνήσουν τα συμβαλλομένα μέρη Βέβαια, στην περίπτωση που επιτευχθεί η συμφωνία. Κρίσιμη ημερομηνία θα είναι το πότε θα μπει στον ΠΟΕ η Ρωσική Ομοσπονδία. Μέχρι τον Ιούλιο του 2012, τότε θα γίνει αυτό. Και τότε θα, θα κρυθεί το τι θα γίνει με τις δεσμεύσεις της Ρωσίας. Θεωρούμε ότι υπάρχει προστασία για τους ε, επενδυτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι θα υπάρξει συνέχιση στην ε, παραγωγή. Θεωρούμε ότι είναι ευμενής μας αυτή η συμφωνία και περιμένω να ακούσω τη γνώμη σας. Σας ευχαριστώ. Ο συνέδριος Τζέρεκ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μεγάλος εξαγωγές αυτοκινήτων και μεγάλος εξαγωγές ανταλλακτικών. Περίπου 9 δισεκατομμύρια ευρώ αξίζουν οι εξαγωγές που κάνουμε προς τη Ρωσία. Υπάρχουν λοιπόν χαμηλή τελωνιακή δασμή και διάφορα, διάφορες απαλλαγές, φοροαπαλλαγές. Υπάρχει ένας κίνδυνος μεταεγκατάστασης επιχειρήσεων. Γι' αυτό η συμφωνία εμπεριέχει μηχανισμούς αποζημίωσης. Έτσι η Ρωσία θα εισάγει ανταλλακτικά από την Ένωση θα μειώσει τελωνιακούς δασμούς σύμφωνα με τον πίνακα 1 και τον πίνακα 2 και θα υπάρχει ένα κατόφλιο το, του 3%. Η συμφωνία επίσης αφορά την περίπτωση κατά την οποία υπάρχει μια μείωση πάνω από 25%. Και έχει μια μεταβατική περίοδο η Ρωσία μέχρι το 2018. Εκεί βλέπετε οι εταιρείες έχουν κρατικές επιχορηγήσεις. Άρα αυτό αυξάνει την ανταγωνιστικότητά τους. Οι Ρώσοι θέλουν να μειώσουν βέβαια την ανεργία τους. Ποιος ξέρει αν αυτή η συμφωνία τελικά θα μας βοηθήσει. Νομίζω ότι είναι καλή συμφωνία για την Ένωση, αλλά πρέπει να την υπογράψουν οι Ρώσοι. Το θέμα είναι, η συμφωνία αφορά μόνο τη Ρωσική Ομοσπονδία ή αφορά Ρωσία, Λευκορωσία, Καζακστάν, τον τελωνιακό αυτό χώρο, την τελωνιακή ένωση αυτή. Το παράρτημα 5 αναφέρεται σε χώρες. Μήπως θα ήταν καλύτερο να λέμε επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ενώσης αντί να αναφέρουμε χώρες. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να διευκρινιστεί. Και κάτι άλλο. Τι, ποια είναι η βάση για το κατόφλιο, το κατόφλιο που αναφέρονται στον πίνακα 3. Λοιπόν, είναι μια, χρειάζεται να ρυθιστούν και διάφορες τεχνικές λεπτομέρειες. Κρίμα που η Ένωση δεν υποστήριξε στις διατυπώσεις της στο σεβασμό των ευρωπαϊκών προδιαγραφών διότι αυτό θα δέσμευε περισσότερο ε, τη διατήρηση της ευρωπαϊκής παραγωγής στην Ευρώπη, να παραμείνει η ευρωπαϊκή παραγωγή στην Ευρώπη, παρά να υπάρχει προσφυγή σε εξωτερικούς ε, προμηθευτές. Ευχαριστώ, δεν υπάρχει άλλο θέλει να μιλήσει, υπάρχει εδώ εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ουχή, ουδής. Αν θέλει ο κ. Ε, να πει κάποια λόγια έτσι ολοκληρώνοντας τη συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Να απαντήσω στον συνάδελφο. Από όσο γνωρίζω, η συμφωνία αυτή αφορά μόνο την ρωσική ομοσπονδία, όχι την ένωση τους ε, με Λευκορωσία και ούτω καθεξής. Αν θέλουμε να αναφερθούμε και στην Ένωση αυτή, θα μπορούσαμε να αναφέρουμε και όσα επιμένει να αναφέρει ο Πούτιν. Ίσως θα μπορούσαμε να το επεκτείνουμε στο μέλλον. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις συνεισφορές σας, θα τις λάβω υπόψη. Πολύ ωφέλιμες για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον συνάδελφο Κόβατς. Και εν τη αυτή περίπτωση οι προθέσμοι για τις τροπολογίες είναι 26 Μαρτίου 12 το μεσημέρι. Πριν σας αποχαιρετήσω να σας δώσω κάποιες πληροφορίες. Πρώτα απ' όλα, συνεδρίαση Δευτέρα το απόγευμα, οι συνεδρίασαν συντονιστές, αποφασίστηκε να ζητηθούν ονόματι, τα ονόματα για την αντιπροσωπεία της Κύπρου. Μιλήσαμε για διάλογο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνάντηση για το ψηφιακό πρόγραμμα 21-22 Ιουνίου. Κάποιες μελέτες θα διοργανωθούν από την αντιπροσωπεία της ΚΟΖΑΚ. Συμμετοχή σε διάσκεψη για την κλιματολογική αλλαγή Δεκέμβριο 2012 και ανατέθηκε έκθεση πρωτοβουλίας για τον οδικό χάρτη για την ενέργεια μέχρι το 2050 στην ομάδα EFT. Η επόμενη συνεδρίαση μας ως Επιτροπή, συνεδρίαση Επιτροπής είναι 23 Απριλίου από τις 3 μέχρι τις 18.30 και 24 Απριλίου από το πρωί και, το πρωί και το απόγευμα. Όμως θα έχουμε και κάποια συνεδρίαση της Επιτροπής μας μαζί με την Επιτροπή Μεταφορών βάση του άρθρου 51 την 3η 27 Απριλίου από τις 3 μέχρι τα 8 και 30 στις Βρυξέλλες όσον αφορά τις διασυνδέσεις, τη διευκόλυνση διασυνδέσεων των μεταφορών στην Ευρώπη. Σας ευχαριστώ για τη συνεργασία σας, για τη δουλειά που κάναμε. Ήταν πολύ έντονες αυτές οι τρεις ημέρες και στο επανειδήν. Γεια σας.